Please. Thank you. So we are Ευχαριστώ. Θα αρχίσουμε την συνεδρίαση. Θα αρχίσουμε με τις ψηφοφορίες για την εκλογή Δευτέρου, Τρίτου ή Δευτερής και Τρίτης Αντιπρόεδρου μετά από το Brexit. Πρώτα απ' όλα, χρειαζόμαστε από τις πολιτικές ομάδες τα ονόματα των αναπληρωτών που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Η γραμματεία δεν έχει ονόματα μέχρι τώρα. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν δύο λεπτά διάλειμμα. Will be even more late. Παρακαλώ λοιπόν, μπορεί το προσωπικό να πάρει τα ονόματα των αναπληρωτών. Ας αρχίσουμε από τους σοσιαλιστές, διότι έχουν ένα κάποιο όνομα για τον δεύτερο αντιπρόεδρο και εμείς με τον τρίτο. Εντάξει, το επόμενο. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος σύμφωνα με την διαδικασία θα πρέπει να έχουμε τα ονόματα των αναπληρωτών. Έτσι μου λέει η γραμματεία. Όχι τους υποψηφίους, τους αναπληρωτές που λαμβάνουν μέρος στην ψηφοφορία. Εντάξει.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 Okay, so I Εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε τη διαδικασία. Θα πρέπει να βεβαιώσουμε ότι έχουμε απαρτία. 21 μέλη. Εύκολα μπορούμε να το διαπιστώσουμε αυτό. Υποψήφοι λοιπόν για την ε, εκλογή του Δευτέρου ή της Δεύτερης Αντιπρόεδρου. Θέλει κάποια πολιτική ομάδα να μας δώσει ονόματα υποψηφίων. Η S&D, σοσιαλιστές, Σίσερ Λουένα. Χωρίς περαιτέρω εξήγηση, έχει όλα τα προσόντα για να γίνει αντιπρόεδρος. Άλλοι υποψήφοι. Θέλω επισήμως συνένεση εκ μέρους συμφωνείτε. Να είστε υποψήφιος. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Διανατάσεως της χειρός, εάν είστε υπέρ, παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, συγχαρητήρια. Προχωρούμε στην επόμενη εκλογή. Τρίτου ή τρίτης αντιπρόεδρου. Υποψήφοι, παρακαλώ. Από το ΕΛΚΑ, τον Ντάν Μουτρεάνου, νέο συνάδελφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά έμπειρο ε, συνάδελφος σε εθνικό επίπεδο. Έχει εργαστεί το Υπουργείο Γεωργία Ακομίας και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι πολύ καλός. Συμφωνείτε συνάδελφε. Ναι, συμφωνώ. Πολύ καλά. Ποιος είναι υπέρ, διατάσεως, πάλι, κατά, αποχές. Είστε ο τρίτος αντιπρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής Περιβάλλοντος και σας συγχαίρω. Okay, so on uh, for human after the agreement found uh, between the Council and μεταξύ ε, των δύο συνομοθετών, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση ευχαριστώ. Εσύ φτάσαμε στο 15. Tout est en ordre. So we are going to resume and then... Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, όποιοι θέλουν να φύγουν ή πρέπει να φύγουν, να το κάνουν. Αρχίζουμε με το επόμενο θέμα της μερίσιας διάταξης. το Παγκόσμιο Σύστημα Συλλογής Δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτα από πλοία. Κύριε Πάλος, ευχαριστώ. Βλέπω ότι υπάρχει κίνηση μεγάλη στην αίθουσα. Όπως ξέρετε, οι περισσότεροι σήμερα παρουσιάζω το σχέδιο έκθεσης ώστε να μπορέσει να η Ευρωπαϊκή Ένωση να ευθυγραμμιστεί το Παγκόσμιο Σύστημα Συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση μαζού από πλοία. Αυτό κατέστη απαραίτητο διότι μετά από την εισαγωγή του MRV, μετά πριν από μερικά χρόνια, αποφασίστηκε ότι πρέπει να υπάρχει ένα διαφορετικό σύστημα και ζητήθηκε από την Επιτροπή να ευθυγραμμιστούν τα δύο συστήματα, την στην έκθεσή μου λοιπόν έχω διευρύνει το πεδίο εφαρμογής που προέβλεπε πρώτος επιτροπής, διότι όλοι στην επιτροπή μας που πάντα είναι στην τοπίδα του τι γίνεται σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει για το θέμα των εκπομπών δεξιού του άνθρωπων κάτι να κάνουμε, όχι μόνο να τις μετράμε, διότι μόνο με το μέτρημα δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε βελτίωση του συστήματος. Αφού λοιπόν υπάρχει τον Νοέμβριο η σχετική ε, δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί επίγουσας ανάγκης και μετά από την ε, κοινοποίηση του Green Deal, του προγράμματος της Επιτροπής που μας παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο, πιστεύω ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται να ενεργήσουμε ώστε να μπορέσουμε για τον τομέα της ναυσιπλοεπίας να κάνουμε κάτι για τον μέτρηση και τον περιορισμό των εκπομπών. Αυτό είναι κάτι το οποίο ελέγχθη σε όλα τα επίπεδα, αναφέρεται και στο Green Deal ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το τομέα της ναυσιπλήμης και είναι μέχρι τώρα μοναδικός τομέας ο οποίος δεν έχει καμία ρύθμιση. Αν δούμε λοιπόν ποια είναι η αναλογία στον τομέα αυτό παγκοσμίω, θα λέγαμε ότι θα μπορούσαμε να τον συγκρίνουμε με την πέμπτη χώρα στον κόσμο με την εκπομπή ε, θερμοκηπίου. Τώρα λοιπόν που έχουμε τα δεδομένα από την MRB που αξιολογήθηκαν για το έτος 2000 και υπολογίστηκαν για το 2018, είδαμε ότι καλύπτονται 10.000 πλοία και όλα αυτά σκάτα την ε, απόπλου και κατά άπλου από τα κοινοτικά λιμάνια ε, ξεπερνούν τις αιτήσια, τα ετήσια επίπεδα του Βελγίου. 130 εκατομμύρια. Θα πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε. Μιλούμε πραγματικά ε, για αριθμούς οι οποίοι είναι πάρα πολύ μεγαλύτεροι από αυτούς που έχουν καταγραφεί όσον αφορά την τον και ίσως αυτό είναι κάτι ε, το οποίο συμβαίνει, η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη από αυτή που έχει καταγραφεί. Δεν είναι πρώτη φορά που μιλούμε για τις ε, εκπομπές στην ευσυπλογία. Το 2013 είχε γίνει και μία αξιολόγηση από την, και εκτίμηση από την Επιτροπή που είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να δούμε τα κατάλληλα μέτρα που θα μας επιτρέπουν να μετριάσουμε. Και στην αξιολόγηση που γίνει επίσης ε, προβλεπόντουσαν κάποια θέματα. Δεν χρειάζεται να ξανακάνουμε όλη αυτή την δουλειά και την αξιολόγηση. Ήδη έχουμε τους αριθμούς από τότε. Και αυτό το οποίο μάθαμε κατά τη διάρκεια της ακρόασης που έγινε τον Ιανουάριο είναι ότι το θέμα της τιμολόγησης δεν θα μας οδηγήσει σε λύση. Δεν θα αποτελέσει λοιπόν κίνητρο ώστε να υπάρχουν πιο αποτελεσματικά πλοία με τη χρήση νέων τεχνολογιών, δεδομένου ότι το ε, κόστος ε, για να αποφύγει κανείς την ε, υψηλή εκπομπή δεν είναι πολύ περισσότερο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε πιο αποδοτικό, καλύτερα ε, λύσεις ανάλογα με, τις, ε, με τα ταξίδια, με τις διαδρομές. Ήδη από το 2008 είχε πει ότι θα πρέπει η αποδοτικότητα να αυξηθεί σε ποσοστά 40% σε κάποια χρόνια, το λάβαμε αυτό υπόψη, αλλά τα μόνα στοιχεία τα οποία πραγματικά είχαμε είναι τα στοιχεία του 2018. Λέμε λοιπόν, και το έχω αναφέρει στην εκθεσή μου, ότι θα πρέπει όντως να έχουμε και πάλι αποδοτικότητα που θα μετρήσουμε από το 2018 έως το 2020. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ε, πλοίων από την ε, εφοπλιστές και από τους υπεύθυνου ότι όντως θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για να βελτιωθεί η τεχνολογία. Με την ε, συμφωνία το Παρισιού είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μία μείωση σίως του 1,5%. Είπαμε ότι θα πρέπει όμως να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι και να μπορέσουμε να, να είμαστε το καλό παράδειγμα για όλους, για μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν εκ μέρους όλων Θα θέλεγα λοιπόν να υπάρξει, ε, αν γίνεται, μεταξύ της MRB και του, αυτά τα οποία ε, λέγει η, IMO, ευθυγράμμιση, θα πρέπει όμως, όπως ακούσαμε και στην ε, ακρόαση, να λέγεται ότι πρόκειται για μία παράμετρο πάρα πολύ σημαντική, διότι μας ζητούν το, όλοι οι υπεύθυνοι να μπορέσουμε να μετρήσουμε το απετύπωμα. Έτσι λοιπόν οι ερευνητές οι οποίοι εργάζονται για το θέμα αυτό θα πρέπει να μας βοηθήσουν. Κατά τρίτον, θα ήθελα να ασχοληθούμε με το μηφέιν, το οποίο είναι το μεθάνιο. Ξέρουμε ότι αυτό το θέμα με απασχολεί πάρα πολύ και με ενδιαφέρει. Θα πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή, να το μελετήσουμε και αυτό το θέμα, όχι να ξέρουμε τι θα γίνει σε 100 χρόνια, αλλά πολύ πιο βραχυπρόθεσμα. Πρόκειται για μία πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση τις εκπομπές μεθανίου να τις μετρήσουμε τώρα, αλλά πρέπει να πω ότι υπάρχουν συγκριτικές αναλύσεις. Άκουσα στο σχετικό εργαστήριο που έκανε πριν από δύο εβδομάδε στο Βερολίνο η Επιτροπή ότι υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τον ε, ε, εξοπλισμό, για τις μεθόδους μέτρησης. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι όλο και περισσότερο μας λένε οι ότι θέλουν να ε, χρησιμοποιούν LNG. Εξαιτία των καλών μετρήσεων της ποιότητας του αέρα. Επίσης, για το θέμα αυτό, μιλήσαμε σε υπεύθυνου των λιμένων, άτομα που ζουν κοντά στα λιμάνια και για αυτούς το αρνητικός αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, που κυρίως οφείλεται στις εκπομπές των πλοίων, είναι πραγματικά ένα θέμα πολύ σημαντικό. Αλλά όπως ξέρουμε όλοι, δεν είμαστε εμείς απόλυτα υπεύθυνοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα είναι υποχρεώσιμο, απλώ από, να ζητήσουμε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση ώστε να μπορέσει στο μέλλον να έχουμε μηδενικές εκπομπές. Και όπως ήδη προανέφερα, ε, θα ήθελα να συμπεριληφθεί και το ΙΤΕΣ. Ο κύριος Τίμεν μας μας το ανέφερε αυτό το θέμα πολλές φορές και αυτό το οποίο θα ήθελα να μπορέσουμε να έχουμε ένα ειδικό ε, ταμείο που θα μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από την χρησιμοποίηση του άνθρακα και να δούμε ποιες θα είναι εναλλακτικέ ε, προτάσεις που θα μπορούσαμε να έχουμε και πηγές ενέργειας ώστε να μπορέσουμε στον τομέα αυτό να κάνουμε κάτι. Βεβαίως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας και κανείς δεν μπορεί να το κάνει μόνος. Θα πρέπει λοιπόν μέλος ε, των ε, κονδυλίων που έχουμε στο ETS να το μεταφέρουμε εδώ και όσον αφορά τους στόχους πρωτικότητας, όπως είπαμε, το μέχρι το 30 θέλουμε να υπάρχει, όπως είπαμε, ε, βελτίωση της τάξης του 40%. Αυτό είναι κάτι που είναι ιδιαίτερα προσφυλές, διότι ίσως οι διάφοροι φοπλιστές δεν θα μπορέσουν να κάνουν μόνοι τους τις απαραίτητες επενδύσεις. Γιατί και σε αυτή την περίπτωση ίσως θα πηγαίνουν πιο αργά τα πράγματα. Αν λοιπόν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι ώστε να υπάρχει καλύτερη τεχνολογία και ως πολιτική να δώσουμε εμείς κάποια στοιχεία, θα βοηθήσουμε την κατάσταση. Διότι και εμείς δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τεχνολογία στον τομέα της ναυσιπλοείας στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Θα δώσω το λόγο στους χιώτες συζητητές, ξεκινώντας με το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια. Ήθελα να επανέλθω στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, όχι για το θέμα του MRV, του ΠΙΕ, e, αλλά υπάρχουν δύο σημεία τα οποία θα ήθελα να εξετάσουμε. Η πρόταση της Κομισιόν αποδυναμώνει την κατάσταση, γιατί δεν μετράμε μόνο το φορτίο αλλά και την χωρητικότητα και αυτό είναι λάθος πιστεύω. Άρα στο σημείο αυτό υποστηρίζω την εισηγήτρια ότι θα πρέπει να μετράμε το πραγματικό φορτίο. Επίσης και το Συμβούλιο είναι υπέρ αυτής της προσέγγισης. Έτσι πρέπει να γίνει λοιπόν. Ε, το ίδιο κάνουμε και με την, ε, τις αεροπορικές μεταφορές. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι πραγματικά μεταφέρεται και όχι τι τεχνικά ε, θα μπορούσε να μεταφερθεί και θα πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο με τον τρόπο αυτό να χρησιμοποιούνται αποδοτικά τα πλοία. Μετά υπάρχει ένα άλλο θέμα που έθιξαν οι συνάδελφοι στην ομάδα μου. Η Κομισιόν απευθύνεται στους πλειοκτήτες, αλλά μερικές φορές δεν είναι οι πλειοκτήτες αυτοί που επηρεάζουν το πώς χρησιμοποιείται στη πράξη ένα σκάφος. Θέλουμε να μιλάμε λοιπόν για operators, δηλαδή για φορείς εκμετάλλευσης των πλοίων, όπως κάνουμε και για τις αεροπορικές μεταφορές. Νομίζω ότι υπάρχει ευρεία συνένεση και για το σημείο αυτό. Μετά υπάρχει ένα αρκετά τολμηρό ε, βήμα ε, όπου προχωρούμε αρκετά πιο μπροστά από την πρόταση της Κομισιόν. Συμφωνώ ότι πρέπει να ενεργήσουμε και να ενεργήσουμε γρήγορα. Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι ο μόνος τομέας όπου δεν εφαρμόζεται νομοθεσία σχετικά με το κλίμα και το περιβάλλον. Είναι καιρός πλέον να ε, δράσουμε και αυτό το τόνισε ήδη η πρόεδρος της Επιτροπής ως μέρος του Green Deal, της Πράσινης Συμφωνίας. Είμαι υπέρ λοιπόν της ε, ταχείας ε, ε, προόδου στο θέμα αυτό. Από τους ψηφοφόρους μας συχνά ακούμε να μας μιλάνε για τις ευθύνες που έχει ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών και πώς πρέπει να είναι υπόλογος. Πώς θα το κάνουμε αυτό για την ομάδα μας και για το Συμβούλιο. Είναι σημαντικό να γίνει μια εκτίμηση αντικτύπου. Ρωτάω λοιπόν την Κομισιόν, η εκτίμηση αντικτύπου που έγινε το 2013 αρκεί ή θα μπορούσε να διευρυνθεί, να γίνει ε, μια ευρύτερη μελέτη ε, αντικτύπου. Ε, αυτό είναι δυνατόν, είναι εφικτό. Φυσικά ε, το μεταξύ μας ολάβησε το Brexit που άλλαξε τις συνθήκες, αλλά δεν νομίζω ότι ε, θα έχει νόημα να μετατοπιστούν οι μεταφορές προς το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να απευθυνθώ προς την εισηγήτρια. Ε, δεν έχει σημασία ε, από πού προέρχεται ή πού καταπλέει το σκάφος, ούτως ή άλλως πρέπει να υπόκειται σε αυτό το καθεστώς. Κοίταξα κάποιους υπολογισμούς και φαίνεται ότι κάτι τέτοιο θα επηρέαζε τις τιμές για τον τελικό καταναλωτή, αλλά σε πολύ μικρό ποσοστό. Ε, θα ήθελα όμως να ρωτήσω για βαριά εμπορεύματα, όπως το τσιμέντο, το σκυρόδεμα, αυτές οι μεταφορές πώς θα επηρεάζονταν από ένα τέτοιο σύστημα. Λοιπόν, το γεγονός ότι θα υπάρξει μικρός αντίκτυπος για τις τιμές σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και αυτές τις μεταφορές ε, στο σύστημα ETS. Ε ε, θα μπορούσαμε έτσι να αποφύγουμε και τη διαρροή άνθρακα. Αλλά όπως για το θέμα του, του τσιμέντου, όπως σας είπα, θα πρέπει να το εξετάσουμε και αυτό το σημείο. Κάτι άλλο. Ακόμα και αν μειώσουμε τις εκπομπές περισσότερο από 30%, πρέπει να φτάσουμε σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Φυσικά θα μπορούσαμε να ε, αυξήσουμε το, να διευρύνουμε το ταμείο αυτό, αλλά αν ε, ε, πρόκειται να έχουμε και διεθνή υποστήριξη για την προσέγγιση αυτή. Θα πρέπει να γίνει διαθέσιμο το Ταμείο και για ε, φορείς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάω από πείρας. Ε, δείτε τι έγινε στον τομέα της ε, αεροπλοείας, όπου ε, το Ταμείο είναι διαθέσιμο μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, εδώ πρέπει να είναι διαθέσιμο και εκτός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ την εισηγητρία για την καλή, πολύ καλή αυτή έκθεση. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι θεωρώ ότι ε, είναι πολύ κοντά στην γραμμή της ομάδας μας αυτό που θέλουμε εμείς να γίνει και ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα βήματα. Το MRV δεν, ε, δεν πρέπει να είναι ένα σύστημα απλώς μέτρησης της κατάστασης αλλά και βελτίωσης της κατάστασης θα ήθελα να αρχίσω κι εγώ όπως και η συγγήτρια ε, λέγοντας, ε, το, ε, λέγοντας πόσο σημαντικός είναι αυτός ο τομέας αλλά βέβαια υπάρχει και μεγάλη δυναμικότητα για το μέλλον του τομέα της ναυσιπλοείας. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη νομοθεσία ώστε να παίξουν το ρόλο που τους αντιστοιχεί στα πλαίσια της Συμφωνίας του Παρισιού θα πρέπει ο τομέας της ναυσιπλοεία να συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης. Όπως έχουν όμως σήμερα τα πράγματα, βλέπουμε το αντίθετο. Βλέπουμε ότι το 2050 μιλάει για αύξηση, κάποιοι μιλάνε για αύξηση 250% των εκπομπών. Αυτός ο κλάδος λοιπόν είναι ένας από, τους, ε, μεγαλύτερους, ε, από τις μεγαλύτερες πηγές ε, εκπομπών παγκοσμίω. Ε, είναι ανάγκη λοιπόν να κάνουμε κάτι περισσότερο ε, και να φροντίσουμε, να εξασφαλίσουμε ότι θα εφαρμόζουμε τα υψηλότερα δυνατά ε, πρότυπα και όχι και να μην ε, στερήσουμε ως προς το Παγκόσμιο Σύστημα Συλλαγής Δεδομένων. Συμφωνώ με τον Πίτερ για το φορτίο. Είναι σημαντικό να μετράμε την πραγματική κατάσταση και όχι κάποιες τεχνικές ιδέες. Και επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα, να θεσπιστούν μέτρα, ούτω ώστε να υπάρχει ένα ανώτατο όριο για το πόσο μπορεί κανείς να εκπέμπει ε, όταν διανύει μια συγκεκριμένη απόσταση. Ε, το να συμπεριληφθεί στο σύστημα MRV. Επίσης, ε, ε, είμαι σύμφωνη για την ε, αναφορά που γίνεται στο σύστημα ETS, στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής. Συμφωνώ με τη σχετική παράγραφο και θα ήθελα και εγώ να ενθαρρύνω το MRV να πιέσει το ETS για τη συμπερίληψη και αυτού του κλάδου. Και χαίρομαι που το ανέφερε αυτό και ο Πίτερ. Νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα του Ταμείου, αλλά δεν θα πρέπει να καθυστερήσουμε υπερβολικά τη συζήτηση αυτή, γιατί τώρα ε, έχουμε ε, την ευκαιρία ανοιχτή μπροστά μας, γιατί και η Κομισιόν βλέπει ότι υπάρχει η σχετική ανάγκη και έτσι θα δώσουμε στον ναυτιλιακό κλάδο μια μοναδική ευκαιρία να βελτιωθεί, να πάρει χρήματα από το σύστημα για να μεταρρυθμιστεί αυτός ο κλάδος. Το MRV λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να ε, καταπολεμήσουμε τις εκπομπές από αυτόν τον κλάδο. Θα ήθελα να καταλήξω με ένα σημείο ε, στο οποίο δεν συμφωνώ και αυτό είναι το σημείο που αφορά τους λιμένες. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε περισσότερα μέτρα από αυτά που προτείνει απλώς η Κομισιόν. Ε, πρέπει να δράσουμε τώρα. Ξέρουμε ότι στα λιμάνια υπάρχουν εκπομπές ε, που ε, είναι σαν μια μικρή χώρα, σαν τη Μάλτα. Ε, δεν μπορεί να δεχτούμε αυτή την κατάσταση να υπάρχουν τέτοιες εκπομπές. Πραγματικά αυτό είναι ε, πολύ επιβλαβές για την υγεία των ανθρώπων που ζουν στα λιμάνια. Πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο στα πλαίσια του MRV για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορώ να δεχτώ το επιχείρημα ότι αυτό αφορά την Επιτροπή Τράνη, την Επιτροπή ή οποιαδήποτε άλλη επιτροπή. Είναι θέμα υγείας των πολιτών και πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω στα πλαίσια του MRV για να μην εκπέμπουν τα ε, πλοία, ενώ βρίσκονται ελιμενισμένα, ε, σταματημένα μέσα στο λιμάνι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια, γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ τεχνικό και η εργασία αυτή ήταν πολύ τεχνική. Ευχαριστούμε λοιπόν για αυτή την εξαιρετική δουλειά που πραγματοποιήθηκε και που υπενθυμίζει τους στόχους πέρα από τις τεχνικές πτυχές, τις φιλοδοξίες που θα πρέπει να έχουμε όσον αφορά την ενεργειακή μετάβαση του ναυτιλιακού κλάδου. Ε, φαίνεται δεν υπάρχει μετάφραση σε κάποιες γλώσσες. Ε, ο πρόεδρος, μπορείς να ξαναρχίσεις ή μάλλον μπορείς να συνεχίσεις, λέει ο πρόεδρος. Οι διερμηνείς ακούνε την ε, σκιώδη εισηγήτρια. Ε, η ελληνική καμπίνα ακούει πάντως. Ωραία. Ε, επαναλαμβάνω. Είναι ένα τεχνικό θέμα λοιπόν να έλεγα, αλλά η συγκεντρία δεν ξεχνάει τους, τις φιλοδοξίες που θα πρέπει να έχουμε στο να εντάξουμε την αυτιλία στα πλαίσια της ενεργειακής μετάβασης. Επίσης κάτι που είναι σημαντικό και το λέει η συγκεντρία, είναι να μην υποχωρήσουμε σε σχέση με τις φιλοδοξίες που έχει θέσει για τον εαυτό της η Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιες και αν είναι οι φιλοδοξίες του IMO. Θα ήθελα να αναφερθώ στα διάφορα σημεία. Όσον αφορά τις εκπομπές, υποστηρίζω την ε, επέκταση των εκπομπών που ε, να μην καλύπτουν μόνο το διοξείδιο του άνθρακα, αλλά όλα τα αέρια του θερμοκηπίου. Και μάλιστα ε, θα έλεγα να μην περιλάβουμε μόνο τα σόξ και τα νόξ, δηλαδή οξύδια του θείου και του αζότου, αλλά ε, γιατί να δημιουργούμε ζώνες χαμηλών εκπομπών και να μην συμπεριλάβουμε και αυτές τις εκπομπές μέσα στην έκθεσή μας. Κατά τη γνώμη μου, ε, λείπει μία εκτίμηση των ε, καυσίμων στο, στους θαλάσσιους βιοτόπους, στη ρήπανση της θάλασσας. Όσον αφορά το ETS, ε, υπεθύμησε η συγκήτρια ότι το 2016 τάχθηκε υπέρ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η πρόεδρος της Επιτροπής το έλαβε αυτό στο Green Deal. Έγινε και μια μελέτη αντικτύπου. Εγώ θα υποστηρίξω τη θέση να περιληφθεί η ναυτιλία στο σύστημα ETS, αλλά με, τρία, με τρεις επιφυλάξεις. Το πρώτο σημείο είναι το Ταμείο Απαλλαγής από τις Εκπομπές ε, ε, που ανέφερε ο συνάδελφος ε, του ΕΛΚ. Η πρόταση αυτή 30% του Ταμείου να προέρχεται από τον αυθυλικό κλάδο μου φαίνεται ότι είναι σημαντικό το 30% είναι λίγο μάλιστα. Θα έλεγα να προτείνουμε κάτι περισσότερο, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι ένα δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο, ενώ οι ανάγκε είναι πολύ μεγαλύτερε. Και μετά σκέφτομαι και κάτι άλλο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μα τι ε, ε, θελοντικέ προσπάθειε που κάνει ο αναφυλιακό κλάδο όσον αφορά την ενεργειακή μετάβαση. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πλειοκτήτε, εφοπλιστέ σήμερα που επενδύουν ήδη και όσον αφορά τον τρόπο πρόωση με και σε ε, χρήση του υδρογόνου. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την μεταβατική περίοδο κατά την οποία θα συνεχίσουν μεν να εκπέμπουν και θα πρέπει άρα να πληρώνουν στα πλαίσια του ETS ενώ ταυτόχρονα ε, ε, και σε θελούσια βάση ακολουθούν μια πολύ θετική στάση. Να, υποστηρίξω, λοιπόν, να υποστηρίξουμε την ε, συμπερίληψη στο ATS, ε αλλά με αυτά τα σημεία. Ε, επίσης, θα προτείνω ε, το εξής. Το λιώνοντας, μία ετικέτα ε, ναυτιλίας που θα πρέπει να αναπτυχθεί μαζί με τις μη κυβερνητικέ οργανώσει και θα πρέπει να περιληφθεί στο ETS. Όσον αφορά τη διαρροή άνθρακα, νομίζω ότι έχει μια πολύ έξυπνη εισηγήτρια που περιλαμβάνει τον ορισμό του ε, λιμανιού όπου κάνει σκάλα το καράβι. Ε, πιάνει σκάλα το καράβι. Νομίζω ότι για τις εκπομπές δεν θα πρέπει να κάνουμε πίσω. Θα πρέπει να διατηρήσουμε τον υποχρεωτικό χαρακτήρα ε, και όσον αφορά ε, τον καθορισμό των προτύπων ενεργειακής απόδοσης, το 40% ναι, η μείωση δηλαδή 40% μέχρι το 2030, ναι, νομίζω ότι είναι ένας δρόμος που μπορούμε να ακολουθήσουμε και επιτρέπει ιδίω στον κλάδο να χρησιμοποιήσει τα μέσα που είναι στη διάθεσή του και ιδίω την μείωση της ταχύτητας όπως είπατε κι εσείς. Ε, συμφωνώ κι εγώ να υποστηρίξουμε ε, την... Ε, ε την, την αλλαγή της ταχύτητας των σκαφών σαν μέσο μάλλον όμως και όχι σαν στόχο. Ε, υπάρχει βέβαια και ε, το Green Deal ε, το λιμάνι της Μασαλίας, παραδείγματο χάρη, να έχει ακολουθήσει ήδη αυτό το δρόμο και θα προτείνω και κάτι άλλο. Οι ε, ποτάμιες μεταφορές ε, όταν γίνονται μεταφορές από την θάλασσα προς τις, ε, ε, την την εσωτερική ναυσιπλοεία. Ε, νομίζω ότι όντως αυτό πρέπει να προσθεθεί και να συμπεριληφθεί και η εσωτερική ναυσιπλοεία. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Ευχαριστούμε. Ζωάλ Μελά έχω στη λίστα μου από την ομάδα ID, αλλά δεν είναι κανείς εδώ. Εντάξει. ECR. Ο κύριος Βοντρά, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα το θετικό σκέλος. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια για την έκθεση. Και για όλες τις προσπάθειες που κατέβαλε για την κατάρτισή της. Υπήρξε πολύ καλή συνεργασία και χαιρετίζουμε και κάποιες ε, νέες πτυχές ε, που εισήχθησαν μέσω των τροπολογιών. Όχι μόνο μια πρόσκληση και έκκληση για περιορισμό του διοικητικού άχθους που είχε ζητήσει το ECR, πάντα είναι κάτι σημαντικό για μας, αλλά και μέτρα ρύθμισης των ε, σκαφών που ρηπαίνουν περισσότερο στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Και να υποχρεώσουμε την, τα σκάφη αυτά να χρησιμοποιούν συγκεκριμένε σύγχρονε τεχνολογίε. Αυτά σίγουρα είναι μέτρα τα οποία στερίζουμε. Από την άλλη, δεν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να καταθέσουμε 34 τροπολογίες για να γίνουν αυτά. Εν γέννη, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτυχάνει μια καλή ισορροπία μεταξύ της απλούστευσης του κανονισμού MRV προκειμένου να υπάρξει συντονισμός με τον ΆΙΜΟ και από την άλλη έχουμε και τη διατήρηση της ακαιρεότητας σε ό,τι έχει να κάνει με την συλλογή πληροφοριών στο ευρωπαϊκό μας σύστημα. Εφόσον το σύστημα του IMO, του Διεθνού Οργανισμού Ναυτιλία, ακόμα δεν έχει κάνει έναν ε, πλήρη κύκλο συλλογική δεδομένων, θα ήταν πρόωρα από εμά να επιμείνουμε στην ευθυγράμμιση ή σε κάποια ουσιαστική τροποποίηση του συστήματος. Μάλιστα, η πλήρης ευθυγράμμιση μεταξύ του ευρωπαϊκού και του συστήματος ε, του IMO ε, θα υπονόμευε τους ε, στόχους της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που έχει ως στόχο την παροχή κινήτρων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και παροχή κινήτρων και ενθάρρυνσης προς τους Φορεί του κλάδου να στραφούν προ πιο φιλικέ προ το περιβάλλον τεχνολογίε. Δεν πρέπει λοιπόν να προκαταλάβουμε την αναθεώρηση τη οδηγία 94 και να επεκτείνουμε το ευρωπαϊκό ε, σύστημα ETS ε προς, ε προς την ναυτιλία χωρίς να μελετήσουμε τον αντίκτυπο ε, της συμπερίληψης όλων των αερίων του και όχι μόνο του διοξιδίου του άνθρακα. Η ομάδα μας λοιπόν θα προτιμούσα να επικεντρωθεί αυτή η πρόταση πρώτον στην ε, σύσταση ενός του συστήματος MRV για την συλλογή των δεδομένων που απαιτούνται για την ε, δημιουργία ενός σημείου αναφοράς πριν προωθήσουμε επιπλέον νομοθεσία για ε, στόχους που έχουν να κάνουν με όλο τον κλάδο σε μια ξεχωριστή πρόταση. Από αυτή την άποψη λοιπόν θα καταθέσουμε μια σειρά τροπολογιών που θα αντικατοπτρίζουν ακριβώ αυτές τις παρατηρήσεις. Thank uh, την Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, είναι η έκθεση πολύ θετική και ένα μεγάλο μπράβο αξίζει στην εισηγήτρια. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται επί της επέκτασης ε, του ETS και έχει στην ευθυλία, αλλά θα μέσα του 2021 προβλέπεται κάτι τέτοιο και αυτό είναι πολύ αργά. Ε, το σχέδιο έκθεση θέλει να συμπεριλάβει την αυτιλία στο σύστημα ETS ε αυτή τη στιγμή. Το εφιστάμενο σύστημα MRV ε απλώ συλλέγει πληροφορίε. Δεν χρειαζόμαστε και άλλα στοιχεία και δεδομένα. Ξέρουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι εκπομπέ από την αυτιλία το σύμμετρο δυνατόν. Ε, συνήθως ε, είμαστε δύσπιστοι προς το ETS γιατί πρόκειται για μια λύση με βάση την αγορά που προς το παρόν δεν έχει θετικά αποτελέσματα. Όμω, σε αυτή την περίπτωση ε, θέλουμε ένα δεσμευτικό στόχο του 40% μείωση μέχρι το 2030. Κάτι το οποίο δεν καλύπτεται στις τροπολογίες προς την πρόταση της Επιτροπής είναι το μέγεθος των σκαφών, των πλοίων. Υπάρχουν διατάξεις του, 2, του άρθρου 2.1 για να έχουμε περισσότερα ε, πλοία. Αντί για 5.000 χωρητικότητα μπορούμε να πάμε στα 4.000. Θα συμπεριληφθούν έτσι 250 πλοία ακόμα. Κάποια θα είναι και πετρελαγωγά. Πετρελοφόρα μάλλον. Ε, στο πεδίο εφαρμογή, σε μια σειρά παραρτημάτων, αναφέρονται κάποια σκάφη τα οποία είναι πάνω από 400 τόνου χωρητικότητα. Ε, ζήτησα από την Τραν για κάποια στοιχεία. Αξιοποιώντα την ε, βάση δεδομένων Clarkson, αν επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογή σε όλα τα σκάφη άνω των 300 τονών, θα συμπεριλάβουμε πάνω από 2.500 ε, ε, πλοία. Και φεριμπότα, αλλά ακόμα και πετρελοφόρα. Υπάρχει απαλλαγή για τα αλλιευτικά. Ίσως πρέπει να εξαιρέσουμε όμως από αυτή την απαλλαγή ε, κάποια είδη αλευτικών σκαφών, τα μεγάλα, τις στράτες, και υπάρχει εξαίρεση και για τα πολεμικά σκάφη. Το Αμερικανικό Ναυτικό, για παράδειγμα, είναι από τους μεγαλύτερους ρηπαντέ στον πλανήτη και δεν νομίζω ότι πρέπει να παρέχουμε τέτοιες απαλλαγέ για τα πολεμικά πλοία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Βάης, ξεκινώντας τη διαδικασία Catch the Eye, η κυρία Νταλή μετά. Άλλος κανείς. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Γιούτα Πάουλους για την έκθεσή της. Η ιδέα αυτή για ένα ταμείο είναι εξαιρετικά θετική. Και τα κίνητρα για το πώς τα κονδύλια του Ταμείου μπορούν να επιστραφούν στον κλάδο για λόγους καινοτομίας και έρευνας. Αυτό είναι μια εξαιρετική ιδέα, ένα εξαιρετικό μέσο και εργαλείο που μπορούμε να αξιοποιήσουμε και σε άλλους τομείς, σε άλλους κλάδους της βιομηχανίας μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι στην έκθεση υπογραμμίζουμε την ε, ε, αξία, την έννοια μάλλον, του φορτίου που μεταφέρεται. Είναι πολύ τεχνικός αυτός ο όρος βέβαια, αλλά είναι σημαντικό για την ε, Επιτροπή μας ε, να ε, δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το σκέλος καθώς προχωράμε στη διαδικασία. Δύο στοιχεία ήθελα να επισημάνω από τακτικής άποψης. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ETS. Όλοι Περιμένουμε με ανυπομονησία ο IMO, το σύστημα του ΟΗΕ δηλαδή, να περάσει προς μία ε, απομάκρυνση από τον άνθρακα για, την, ε, τον κλάδο ευρύτερα. Αλλά εμένα με προβληματίζει, από πλευράς τακτικής και πάλι, ότι μπορεί να αποτύχουμε εάν αυτή τη στιγμή επιμείνουμε για τον, για τον επόμενο χρόνο. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα μπορέσει να αποδείξει ότι μπορεί να πετύχει μια συμφωνία σε επίπεδο IMO. Γιατί αν συμφωνήσουμε επί αυτού του συγκεκριμένου ζητήματος, τελικά μπορεί να αποτύχουμε στον απότερο μας στόχο, που είναι να έχουμε όλη την παγκόσμια ναυτιλία και όχι μόνο το ενέκτο αυτής. Είναι θέμα τακτικής λοιπόν. Γιατί μπορεί τώρα να ασκήσουμε πολύ μεγάλη πίεση αυτή τη στιγμή, μετά να κάνουμε πίσω και να μην έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για του Ευρωπαίους πολίτες. Άλλο ζήτημα. Η baseline, το σημείο αναφοράς που αναφέρεται στην νετροπολογία τροπολογία 27. Ε, κατανοώ τα επιχειρήματά σας αλλά ο στόχος μείωσης των εκπομπών κατά 40% μέχρι το 2030 όπως έχουν υιοθετηθεί από τον IMO αυτή τη στιγμή, βασίζονται σε στοιχεία του 2008. Αν πούμε, αν, αν πούμε εμείς 2018, αυτό απευθύνει ένα σφαλμένο μήνυμα προς τους ε, προτεργάτες ε, του κλάδου αυτού, όπου έχουμε φορείς, εταιρείε, έχουμε δει ότι έχει κάνει μέρες, ας πούμε, που ήδη έχουν κάνει κινήσεις ε, απομάκρυνσης από τον άνθρακα και αποτελούν ένα παράδειγμα προς τον ευρύτερο κλάδο ότι μπορούν να στραφούν σε άλλα μέσα και τεχνολογίες πιο φιλικές προς το περιβάλλον ε, με έναν βιώσιμο τρόπο. Αν λοιπόν μεταφερθούμε εμείς σε στοιχεία του 2018, στην ουσία ε, λειτουργούμε τιμωρητικά προς αυτούς που έδωσαν το καλό παράδειγμα. Και πάλι από πλευρά τακτική, ε, το αναφέρω. Θέλουμε όντως να τιμωρήσουμε τους προτεργάτες, τους πρωτοπόρου σε κάθε κλάδο. Γιατί μετά κανένας δεν θα θέλει να αναλάβει αυτό το ρίσκο ε, και να προβεί σε μέτρα τομή σε σχέση με αυτά που ακολουθούν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ευχαριστώ κύριε Ανταλή, ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια θα ήθελα να σταθώ σε κάτι που αναφέρθηκε μόλι, γιατί εμεί εξετάζουμε το θέμα των εκπομπών τη ναυτιλία εδώ και πολύ καιρό. Από τη στρατηγική του 2013, για παράδειγμα, μιλούσαμε για μια σταδιακή ενσωμάτωση των εκπομπών της ναυτιλίας στους ευρύτερους στόχους ε, μείωση των εκπομπών αερών του θερμοκηπίου και τα πράγματα δεν έχουν κινηθεί όσο γρήγορα θα θέλαμε. Και τελικά είχαμε πολύ μικρή πρόοδο. Πού φτάνουμε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση όπου περιμένουμε από τον IMO να αναλάβει δράση, δεν το κάνει όμως. Ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι κλάδοι συμβάλλουν στο στόχο τη ε, ε, απομάκρυνση από τον άνθρακα. Αυτό πρέπει να κάνει και η ναυτιλία. Τώρα έχει θεσπιστεί λοιπόν το σύστημα MRV, αλλά ακόμα και η τρέχουσα πρόταση τη Επιτροπή νομίζω ότι δεν θέτει καθόλου δεσμευτικού στόχου μείωση, ούτε μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων για τον τομέα της ναυτιλίας. Χρειαζόμαστε ένα ε, μείγμα λοιπόν μέτρων που θα είναι και βραχή και μάχρο πρόθεσμα. Το Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, ζητά την ε, επέκταση του συστήματος ETS ε και στον τομέα της ναυτιλίας και ακούσαμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θέλει να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Η επέκταση του EU ETS ε στην ναυτιλία και στις μεταφορές μπορεί να βασιστεί και στο ισχύον πεδίο εφαρμογής του κανονισμού MRV. Εγώ πιστεύω σε ισχυρά μέτρα, παρότι τα νέα μέτρα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και την διεθνή ανταγωνιστικότητα των σκαφών με ευρωπαϊκή σημαία και να μην δημιουργούν ε, διπλή νομοθεσία για τον κλάδο. Αναφέρθηκαν και οι καθαροί λιμένε και η Μάλτα πιο συγκεκριμένα. Εγώ επισημαίνω και πάλι πόσο αναγκαίο είναι να επενδύσουμε σε καθαρότερου λιμένε. Γιατί τελικά έχουμε Ευρωπαίου πολίτε που μένουν εκεί και θα πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία του. Στηρίζω τη θέση τη συγγήτρια ότι η στόχη μείωση των εκπομπών τη ναυτιλία θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον νέο στόχο για το 2030 και με το στόχο τη ενεργ... κλιματική Και σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να προωθήσουμε και του ε, μηδενικών εκπομπών και τελικά όλο ο κλάδο ναυτιλία να κινηθεί προ την κατεύθυνση των μηδενικών εκπομπών, κατανοώντα αυτό που είπε η συγγήτρια, ότι ε, θέλουμε και τα μέτρα που δεν είναι επαχθή οικονομικά. Σίγουρα χρειαζόμαστε σημαντικέ επενδύσει στην έρευνα και καινοτομία και στήριξη για την ανάπτυξη βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων, το refueling και υποδομέ ε, επαναφόρτηση στου λιμένε μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καθότι πρόεδρος έχω και το προνόμιο να βάζω το όνομά μου στον κατάλογο μελητών. Για την τροπολογία 23 ήθελα να ρωτήσω πώς βλέπετε αυτόν τον μηχανισμό για την αποφυγή της ε, ε, μεταφοράς της φόρτωσης σε άλλους λιμένες. Στην Τουρκία, για παράδειγμα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς βλέπετε να δουλεύει αυτό το σύστημα. Εμείς μπορούμε να το αποφύγουμε, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε την ύπαρξη ενός σωστού και ορθού συστήματος. Ποια είναι λοιπόν συγκεκριμένα η πρότασή σας. Uh, να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε κάτι άλλο εσείς να προσθέσετε. Ωραία. Κυρία Λεωράνς Γκράφ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Ευχαριστώ και την κυρία Συγήτρια. Σας ευχαριστώ για το προσχέδιο έκθεσης. Με τα χαρά ξεκινούμε τις εργασίες ε, και τη συνεργασία μας για αυτό το φάκελο. Ελπίζουμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στο εγγύς ε, μέλλον, εφόσον και το Συμβούλιο πλέον είναι σε θέση να προχωρήσει. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε την ε, πρόταση πέρυσι, σχεδόν πριν από ένα χρόνο, ε, λαμβάνοντας ε, επαρκώς υπόψη τα όσα έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο IMO για ένα σύστημα συλλογής δεδομένων σύμφωνα και με τις διατάξεις περί αναθεώρησης στον κανονισμό μας. βασικός στόχος ε, ήταν ε, η προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας μέσω τεχνικών ε, τροποποιήσεων για να επιτρέψουμε μια σωστή εφαρμογή του κανονισμού από κοινού και με το σύστημα MRV και έτσι να ελαχιστοποιήσουμε το διοικητικό άχθος. Από την άλλη, δεν θέλουμε και να επανομεύσουμε κατά οποιονδήποτε τρόπο τους στόχους του κανονισμού. Εμείς θέλουμε μια σωστή και εύρωστη ε, διαδικασία συλλογής δεδομένων, ε, διαφάνεια, που ήταν βασικό στόχος του κανονισμού, και παροχή κινήτρων για την μείωση των εκπομπών διεξουδίου του άνθρακα. Η πρώτη υποβολή εκθέσεων έγινε το 2018, η πρώτη συλλογή δεδομένων έγινε πέρυσι και είχαμε και μία μάλλον περιμένουμε αυτή τη στιγμή, προετοιμάζουμε στην Επιτροπή μία αναλυτική έκθεση την οποία θα μοιραστούμε μαζί σας στο μέλλον. Έχουμε λοιπόν εύρωστα και σωστά στοιχεία για ένα εντυπωσιακό αριθμό σκαφών ε, που ελιμενίζονται σε ευρωπαϊκούς λιμένες. Θέλουμε να προετοιμαστούμε για τα επόμενα βήματα πολιτικής που, έχουμε, που είχαμε μάλλον εντοπίσει το 2013 στην Στρατηγική της Επιτροπής. Όπως ξέρετε έχουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νέα πολιτική όθηση με την Πράσινη Συμφωνία και δέσμευση για βελτιωμένε κλιματικέ ενέργειε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλου του κλάδου της ευρωπαϊκή οικονομία. Σύμφωνα πάντα και με το πνεύμα τη ε, Συμφωνία του Παρισιού. Η ναυτιλία ως κλάδος είχε μείνει εκτός, όπως είπατε και εσεί από αυτές τι ενέργειε ε, μετριασμού της κλιματική αλλαγή μέχρι τώρα. Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί, ιδίω καθότι έχουμε σημαντικές δυνατότητες ε, μείωσης των εκπομπών σε αυτόν τον κλάδο. Και βέβαια το ETS είναι κάτι το οποίο έχει προταθεί ως μέτρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε ξεκινήσει τις ενέργειές μας στο πλαίσιο ενός, μιας ευρύτερης δέσμης ε, μέτρων που εντάσσονται στην Πράσινη Συμφωνία και σε μια ευρύτερη δέσμη μέτρων που αφορά την αυτιλία. Ορισμένοι αναφέρθηκαν στην προηγούμενη μελέτη αντικτύπου που έγινε το 2013. Πράγματι, θα βασιστούμε σε αυτήν. Ε, το να πούμε ότι αρκεί για την επερχόμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ETS, ε δεν θα το έλεγα αυτό. Θα πρέπει να ε, επαναξιολογήσουμε την κατάσταση υπό το φως αυτής της ενισχυμένης κλιματικής ενέργειας. Αν πάμε σε ένα στόχο 50-55% θα πρέπει να το εξετάσουμε βέβαια. Θέλουμε να θίξουμε το ζήτημα της ναυτιλίας ε, στο ETS ε και τι αντίκτυπο θα έχει σε άλλους κλάδους. Το αν θα έχουμε ανοιχτό κλειστό σύστημα ETS ε προφανώς και θα επηρεάσει και άλλους τομείς. Και βέβαια πρέπει να πάρουμε υπόψη και τον αντίκτυπο του Brexit. Από πλευράς μας λοιπόν ε, θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη για ε, νέα ή πιο επεξεργασμένη μελέτη αντικτύπου. Τώρα, ορισμένα σχόλια εν συντομία για παρατηρήσεις που κάνατε εσείς σε ό,τι έχει να κάνει με το πεδίο εφαρμογή. Αν πρέπει να περιοριστούμε στο διεξουδίο του άνθρακα ή πρέπει να κινηθούμε ευρύτερα προς ε, τα αέρια του θερμοκηπίου η Επιτροπή αρχικά είχε αποφασίσει να επικεντρωθεί στο διοξείδιο του άνθρακα γιατί είναι πάνω από το 95% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκαλεί η ναυτιλία. Αυτό είναι το σκεπτικό μας. Το ίδιο ίσχυε και για το μέγεθος των πλοίων, γιατί με το σημερινό όριο κατόφλι ε, καλύπτουμε το 90% των εκπομπών. Για το φορτίο σημειώνω τη θέση σας Σημειώνω επίση ότι ήταν και η θέση του Συμβουλίου. Θα το σκεφτούμε λοιπόν αυτό. Για τα επιχειρησιακά πρότυπα διεξοδίου του άνθρακα πάλι κατανοώ το επιχείρημα. Είναι κάτι το οποίο συζητείται εκτενώς και στον IMO ε, φέτος. Στην επόμενη MEPC σίγουρα θα μας απασχολήσει το Μάρτιο αλλά και στην επόμενη, τον, το φθινόπωρο. Για το οικονομικό σκέλος, όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να βρούμε επιπλέον χρηματοδότηση για να υποστηρίξουμε αυτή την στροφή του κλάδου, μακριά από τον άνθρακα. Με το ETS σίγουρα τα έσοδα θα μπορέσουν να συμβάλλουν σε αυτή τη χρηματοδότηση και επένδυση σε νέες τεχνολογίες, στην ε, αναδρομική εφαρμογή, retrofitting και ούτω καθεξής. Αυτά από πλευρά μας προς το παρόν. Ευχαριστώ. Η συγγήτρια. Ε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους ε, σκιώδεις συζητητές, με τους οποίους έχουμε πραγματικά μια πολύ επικοδοματική ανταλλαγή απόψεων πριν την κατάρτιση της έκθεσης και για τα όσα είπατε σήμερα. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το όριο των τριών λεπτών, αλλά είναι αρκετά τα ζητήματα που θίξατε. Πρώτον, προς τον Πίτερ Λίζε, είπατε ότι θα πρέπει να είναι ουδέτερα τα μέτρα προς ε, τις ε, πλειοκτήτριες εταιρείε και προς τις χώρες ε, κράτους σημαία. Αυτό ισχύει και από τον MRV και από αυτόν τον κανονισμό, ανεξάρτητα λοιπόν από το κράτος σημαία και από την πλειοκτήτρια εταιρεία αυτό που μας αφορά είναι ποιος μπαίνει στο λιμάνι. Αυτό καλύπτεται από τον κανονισμό. Μπορούμε να μιλήσουμε για το ποσοστό που θα πρέπει να πάει στο ταμείο. Βεβαίω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σίγουρα μπορούμε να βρούμε, να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο ε, να ανοίξουμε το ταμείο προς ε, άλλες εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν είστε κάπου για διακοπές και ε, πληρώσετε κάποιο φόρο στα τρόφιμα που αγοράζετε, δεν θα δείτε έσοδα από αυτό. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να ισχύει και σε εμά, αλλά εντάξει, ξέρω ότι έχετε μεγάλη εμπειρία στι αεροπορικέ μεταφορές. Ναι, βεβαίως, μπορούμε να ζητήσουμε το θέμα των λιμένων μηδενικών εκπομπών. Θα ήθελα ε, να ασχοληθούμε με το ζήτημα της υγείας των πολιτών που μένουν ε, κοντά στα λιμάνια. Για τα οξύδια του θείου και του αζότου και τις σχετικές εκπομπές, πολύ σημαντικό το ζήτημα. Σε σχέση με το διοξίδιο του άνθρακα, το πρόβλημα με αυτά είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να μετρηθούν. Στο διοξίδιο του άνθρακα είναι πολύ εύκολο να υπάρξει μέτρηση το καύσιμο που εισάγεται τελικά θα οδηγήσει σε εκπομπές με, ε, του διοξιδίου του άνθρακα. Όμως με τα οξύδια θείου και αζότου τα πράγματα αλλάζουν γιατί έχουν να κάνουν και με τον τρόπο λειτουργίας της μηχανής, του κινητήρα. Αλλά σίγουρα μπορούμε να καταλήξουμε και εδώ σε μια σωστή προσέγγιση. Κύριε Βάντρο, αν είχαμε ε, άπλετο χρόνο θα συμφωνούσα μαζί σας να περιμένουμε ακόμα 3-5-6 χρόνια, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Εγώ δούλευα παλιότερα σε ένα νοσοκομείο σε ό,τι αφορά την ποιότητα, διαχείριση ποιότητα και είχαμε πολλά έτσι ωραία προγράμματα για το πώ να αντιμετωπίζουμε ασθενεί με συγκεκριμένε νόσου. Κάποιε φορέ όμω οι ασθενεί δεν ακολουθούσαν τα σχέδια αυτά, τα προγράμματα. Επομένω, η κατάστασή του άλλαζε προ το χειρότερο. Και έπρεπε να αλλάξουμε το αρχικό μας πλάνο για να σώσουμε τη ζωή του ασθενούς. Αυτό ισχύει και στη σημερινή κατάσταση. Προς τον κύριο Βόλας. Ε, ναι, συζητήσαμε το πόσες εκπομπές θα μπορούσαμε να καλύψουμε με την επέκταση, διεύρυνση του πεδίου γιατί ήδη καλύπτεται το 9% των ε, εκπομπών από τον υφιστάμενο οικονομισμό. Προτείνω λοιπόν, αν υπάρχει, αν έχετε μια ευρύτερη εικόνα για τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε κάθε συγκεκριμένο κλάδο, μπορούμε να το συζητήσουμε. Για τα στρατιωτικά. Ο Αμερικανικός στρατός από το 2001 έχει εκπέμψει 1,2 εκατομμύρια κυβικούς τόνους ε, εκπομπών. Ναι, αλλά αυτό δεν αφορά ευρωπαϊκά λιμάνια στο σύνολό του. Πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό. Πενίλ, είπατε ότι πρέπει να σκεφτούμε αν είναι συνετό να πιέσουμε τον IMO. Ε, μου έχουν πει ότι μόνο υποπίεση κάνει οποιαδήποτε κίνηση ο IMO. Αλλιώς δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Ε, ενδεχομένως να διαφωνούμε ε, ως προς αυτό, αλλά εγώ πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να ε, πιέσουμε τον IMO και να δείξουμε ότι δεν μπορούμε πια έτσι να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Ε, με τα χαράς να ε, αρχίζουν και αυτοί να εφαρμόζουν το δικό μας σύστημα, το ETS. Κανένα πρόβλημα. Για το δεύτερο σκέλος, για την αλλαγή του σημείου αναφοράς, αν αυτό θα λειτουργούσε τιμωρητικά προς τους πρωτοπόρους. Εμείς κοιτάμε την μέση κατανάλωση, επομένως, η πρωτοπόροι ήδη έχουν επιβραβευθεί γιατί πρέπει να κάνουν λιγότερα για να πετύχουν τον τελικό στόχο του 40% μέχρι το 2030, εφόσον ήδη έχουν φτάσει το 25% σήμερα. Αν είναι 25% κάτω από τον μέσο όρο σήμερα, τους απομένει μόνο ένα 15% για να φτάσουν το στόχο μέχρι το 2030. Επομένως δεν τιμωρούνται με κάποιον τρόπο. Μίρια Μντάλη, σε ευχαριστώ για την υποστήριξη. Χαίρομαι που σου άρεσε η έκθεσή μου. Πασκάλ, το θέμα της ε, διαρροής ε, διοξιδίου του άνθρακα στην δημόσια ακρόαση, νομίζω ότι κατέστη σαφές ότι ε, χάνουμε χρόνο με αυτές τις παρακάμψεις, το επιπρόσθετο κόστος των καυσίμων. Είναι πολύ μεγαλύτερο αυτό το κόστος, λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό ETS θα έπρεπε να υπάρχει το, το ETS να κοστίζει εκατοντάδες ευρώ για να σκεφτούμε το ζήτημα της διαρροής ε, άνθρακα. Δεν νομίζω ότι θα αυξηθούν τόσο πολύ τιμέ στο ETS τα επόμενα πέντε χρόνια τουλάχιστον. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας ευχαριστώ πολύ που μας ε, βοηθήσατε στα τεχνικά ζητήματα. Ήδη είπατε ότι έχει ξεκινήσει η προσπάθειά σας για το ETS, χαίρομαι. Είπατε ότι πρέπει να σκεφτούμε αν θέλουμε ανοιχτό ή κλειστό ETS. Νομίζω ότι η αποφυγή κόστους διαφέρει πολύ εδώ σε σχέση με άλλους κλάδους. Θα ήταν καλό λοιπόν να έχουμε ένα ξεχωριστό ETS αυτή τη στιγμή τουλάχιστον και να σκεφτούμε την ευθυγράμμιση για αργότερα. Εγώ διατήρησα ανοιχτό αυτό το ζήτημα στην πρότασή μου, γιατί θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει ποιο μέτρο είναι καλύτερο και τι πλεονεκτήματα και τι μειονεκτήματα έχει κάθε λύση. Σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες τροπολογίες για τις οποίες θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 11 στην ΕΜΒΗ ψηφοφορία το Μάιο και στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Πολύ ωραία. Και τώρα θα προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Δίνω την προεδρία στην κυρία Αλβίνα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Εγώ είμαι εμπειρογνώμενο σε θέατα αεροπλοίας. Το μεγάλο ποσοστό των δικών μας αεροπλάνων, λιγότερο αποτελεσματικά από αυτά τον είπα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη όταν μιλούμε για μείωση των εκπομπών εξή του άνθρωπου. Continuamos con el punto 16. Αρχίσουμε με το σημείο 16. Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και το αεριοποιημένο καπνό. Πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο μέρους της Γενικής Διάθεσης Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Αντρέη Ρης Για 10 λεπτά του δίνω το λόγο. Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι σας. Ευχαριστώ που κάνετε εδώ αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση. Θα αρχίσω με μία μικρή παρουσίαση για την κατάσταση των πραγμάτων σήμερα όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τον αεροποιημένο καπνό. Λοιπόν, εάν θυμάστε, η σχετική οδηγία άρχισε να εφαρμόζεται από το 2014 η TDC και αφορά όλα τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, το άτμιδα και τα αεροπηρημένα ταπνό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το εξής. Πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε την ελκυστικότητα του καπνού στα νέα. Πρώτα απ' όλα είχαμε την πρώτη ε, νομοθεσία για την ε, μπορέσουμε να ρυθμίσουμε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε κυρίως για τους νέους να εξασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο πρόσπισης της υγείας τους. Είναι θέμα δημόσιας υγείας. Ναι, είμαι εδώ μπροστά. Γι' αυτή αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε κάποια ρύθμιση. Η υπήρχε η σχετική οδηγία και είπαμε ότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε τα πράγματα δεδομένου ότι στην, ε, ε, Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πολλές κείμενες διαφορετικές νομοθεσίες. Θέλουμε, να, θελήσαμε λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε μια κάποια εναρμόνιση. Επίσης, πρέπει να πω ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το πρόβλημα δημόσιας υγείας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί βλέπετε ότι υπάρχουν προβλήματα που μας απασχολούν όπως παραπληροφόρηση, ε, επιπτώσεις ε, ε, μακρυπρόθεσμα και άλλα θέματα τα οποία μας απασχολούν και θέλουμε να υιοθετήσουμε αυτή την προσέγγιση της ρύθμισης. Πρώτα απ' όλα, γιατί στρέφονται στο ηλεκτρονικό τσιγάρο και γιατί εθίζονται κυρίως σύμφωνα με τις Μελέτες του Ευρωβαρομέτρου του 2017. 15% προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό τσιγάρο. 25% ήταν ε, νέοι 15 με 24 ετών που χρησιμοποίησαν το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμφανίστηκε και στις Ηνωμένε Πολιτείες και είδαμε ότι μειώθηκε η κατανάλωση τσιγάρου την τελευταία δεκαετία, αλλά είδαμε ότι τώρα πάρα πολλοί μαθητέ του γυμνασίου προστρέχουν στο άτμισμα. Ξέρω ότι πολλούς από εσάς σας απασχολεί το θέμα της ασφάλειας του ατμήματος. Είδαμε πριν από κάποιους μήνες να υπάρχει πρόβλημα σοβαρό στη ΣΥΠΑ, δεδομένου ότι δημιουργήθηκαν κάποιοι, κατέληξαν σε θάνατο κάποιοι χρήστες. Έτσι λοιπόν υπάρξει αυτή η ανησυχία. Τι κάνουμε για να ρυθμίσουμε την όλη κατάσταση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Προσπαθούμε να παρακολουθούμε εκ του σύναγκες τι γίνεται. Ξέρουμε ότι υπάρχει η σχετική ε, νομοθεσία για τον καπνό. Ξέρουμε ότι χρησιμοποιούνται ε, διάφορα πρόσθετα βιταμινούχα τα οποία θέλουμε να απαγορευθούν και άλλα ε, συστατικά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν εθισμό. Επίσης θέλουμε να υπάρχει ε, μείωση της νικοτίνης και της συγκέντρωσης νικοτίνης όχι πάνω από 20 μικρογραμμάρια μιλιγκράμμ ανά Στην ε, οδηγία δεν γίνεται εναρμόνιση όλων των πτυχών. Πολλά μάθαμε πέρσι. Επίσης, το CBD είναι κάτι που δεν έχει ρυθμιστεί. Συνεχίζουν είναι ελκυστικά όμως αυτά τα προϊόντα μεταξύ των νέων η επιτυχία τους οφείλεται στα διαφορετικά αρώματα που είναι διαθέσιμα. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να απαγορεύσουν τη χρησιμοποίηση τέτοιου είδου αρωμάτων. Ένα είδο, κράτος μέλος ήδη το έχει επιτύχει, οι άλλοι το σκέφτονται. Επίσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, κάνουν ε, διάφορες καμπάνιες ευαισθητοποίησης, να δώσουν τις κατάλληλες πληροφορίες βασιζόμενες στις διάφορες αναφορές και έρευνες που έχουν γίνει και είπα κι αλλού. Τώρα, όσον αφορά τα να αεριοποιημένο καπνό και όλα αυτά τα προϊόντα. Στο TPD υπάρχουν διάφορες διατάξεις για την ρύθμιση αυτών των οποίων ονομάζουμε νέα ε, καπνικά προϊόντα. Όπως ίσως γνωρίζετε, φέτος το Μάιο θα τεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας οδηγίας η απαγόρευση πώληση τέτοιου είδους προϊόντων. Το αεροποιημένο καπνός τι είναι. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες στην αγορά, γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Υπουργή προσπαθεί σύμφωνα με επιστημονικές πληροφορίες να δει πώς έχει κατάσταση. Είδαμε ότι υπάρχουν και διάφορα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες τα οποία προστίθενται εδώ και ε, διάφορα συσκευές που χρησιμοποιούνται. Τα προϊόντα και οι συσκευές αυτές δεν είναι πάντα ε, ρυθμισμένες και έτσι πολλές φορές εκθέτουν ακόμη και τα μικρά παιδιά. Επίσης υπάρχουν διάφορα παραπληντικά μηνύματα τα οποία έχουν εμφανιστεί και λένε ότι αυτά τα προϊόντα είναι εναλλακτικέ λύσεις πολύ καλύτερες από το κάπνισμα, το κλασικό. Πέρσι στην FCTC COP8 λήφθησαν αποφάσεις ώστε να συσταθεί σε όλα τα μέλη να εφαρμόσουν ρυθμιστικά μέτρα τα οποία θα ήταν τα καλύτερα. Εφέτος, στην Ολλανδία, στην COP9, είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός όλων αυτών, ώστε να μην υπάρχει ε, καταστρατήγηση όλων αυτών των διατάξεων πρέπει να εφαρμόζονται τά. Ας δούμε τι ακριβώς έχει γίνει στην Επιτροπή και τι προσπαθούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα αυτό το φαινόμενο. Αν θυμάστε, στην οδηγία ζητάει η Επιτροπή να γίνεται αναφορά στο, να γίνει αναφορά στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο το Μάιο του 2021. Είμαστε σε προπαρασκευαστική φάση και μπορείτε να δείτε ποια είναι τα θέματα τα οποία θα πρέπει να αξιολογήσουμε για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, για τα νέα προϊόντα, για τα, ε, ε, τα υγρό αναπλήρωση, το τι ακριβώς γίνεται με όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία εμφανίζονται στην αγορά. Προσπαθούμε λοιπόν από τις διάφορες πηγές ενημέρωσης που έχουμε στα πλαίσια των ομάδων εμπειρογνωμόνων από τα κράτη-μέλη και με τις ε, ε συντονισμένες δράσεις που αναλαμβάνουμε, να δούμε τι γίνεται επίσης, ζητούμε την άποψη των εμπειρογνωμόνων, γίνονται έρευνες για να δούμε τι ακριβ, περί ακριβώς πρόκειται με όλα αυτά τα προϊόντα, ηλεκτρονικά τσιγάρα και τον αεροποιημένο καπνό. Επίσης πρέπει να γίνει, έχουμε την ε, επιστημονική αξιολόγηση της ΣΕΡ που είναι επιστημονική επιτροπή για θέματα υγείας, περιβάλλοντος και αναδιο εμφανιζόμενων ε, κινδύνων που θα κάνει τις σχετικές της ε, εκθέσεις και επιστημονικές ε, γνωμοδοτήσεις για τα θέματα υγείας που προκύπτουν από την χρησιμοποίηση αυτών των προϊόντων. Έχει γίνει ο σχεδιασμός, το σχέδιο γνωμοδότησης και η δημόσια διαβούλευση θα γίνουν φέτος στην Άνοιξη και η τελική γνωμοδότηση παρουσιαστεί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο φέτος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρης. Έχει τώρα το λόγο πρώτα απ' όλα η κυρία Μανίτς. Um, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πάρα πολύ χρήσιμη παρουσίαση της παρούσας κατάστασης. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις και όλοι ξέρουμε τι ακριβώς έγινε στη ΣΥΠΑ. Γι' αυτό καλό είναι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Ε, έχει ασχοληθεί με το θέμα, αλλά όχι πλήρως. Μία από τις στατιστικές που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες από την ε, ε, παρουσίαση ήταν το άτμισμα εκ μέρους των νέων παιδιών. Ίσως έχετε αυτές τις προφορίες. Θα πρέπει να ξέρουμε αν πραγματικά είναι η πρώτη τους εμπειρία. Δηλαδή δεν έχουν ποτέ καπνίσει πριν, αλλά άρχισαν με το άτμισμα, διότι είναι κάτι το οποίο είναι πιο αποδοκτό σήμερα. Θα ήταν ενδιαφέρον να ξέρουμε αν έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτό το οποίο έγινε στη ΣΥΠΑ ήταν πάρα πολύ ανησυχητικό. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποια ε, θέματα στην οδηγία, τα οποία είναι θέματα αρμοδιότητας των κρατών μελών και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε καλύτερη εναρμόνιση για θέματα όπως το CBD, τα αρώματα, τα πρόσθετα. Πρέπει Λοιπόν, να τοποθετηθούμε δεδομένου ότι έχουμε κάποιες υποφορίες επί του θέματος ή για οποιαδήποτε άλλα θέματα βάσει των μαρτυριών που έχουμε όσον αφορά την ε, ε, πρακτική των καταναλωτών, ώστε να κάνουμε κάποιες αλλαγές στο, θέματα, στο θέμα του ατμήματος. Ίσως αυτό το συμπεριλάβουμε στην έκθεσή μας του χρόνου. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πόσο γρήγορα συνέβησαν τα πάντα εν, μία νυχτή. Και πρόκειται για ένα θέμα το οποίο και πάλι ανήκει στις εταιρείε ε, ε, των οι οποίες θέλουν να διαφοροποιήσουν, που προϊόν τον καπνό, τα προϊόντα και θέλουν να διαφοροποιήσουν τα τα, την παραγωγή τους. Ξέρουμε Επίσης ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύσουμε τις εγγύους. Να μην καπνίζουν, αλλά όχι και να τους προτείνουμε ως εναλλακτική λύση το άτμισμα. Η συζήτηση και η παρουσίαση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Πιστεύω ότι θα πρέπει εκ του σύνταξη να παρακολουθούμε τι γίνεται επί τόπου. Διότι κανένας ε, δεν είχε προβλέψει ότι 20% των νέων θα ε, χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τσιγάρο. Είναι πολύ ψηλό αυτό το ποσοστό και ξέρουμε ποιο είναι ο αντίκτυπο σε όλου του τομεί τη κοινωνία. Υπάρχουν λοιπόν ασαφή θέματα και ξέρουμε ε, πόσο το θέμα των ε, αρωμάτων μπορεί να εθίσει τους νέους. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε τι γίνεται, να δούμε τι γίνεται και επί τόπου από τον καθένα για να κάνουμε την δική μας αξιολόγηση. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά, αλλά τέτοιου είδους πληροφορίες για το τι γίνεται σε κάθε χώρα θα πρέπει να έχουμε το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λίζε τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και να υποβάλω μια ερώτηση. Τι συνέβη στις Ηνωμένε Πολιτείε. Πρόκειται για ένα ερώτημα που πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες θέτουν και δεν μπορέσαμε στην τελευταία διαβούλευση να απαντήσουμε στην Γενική Διεύθυνση Υγείας θα πρέπει να γνωρίζουν οι συνάδελφοι τι ακριβώς συνέβη. Γιατί τόσα άτομα υπέστησαν βλάβες σοβαρές από το ηλεκτρονικό ε, τσιγάρο. Μας προστατεύει εμάς η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ώστε να μην έχουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Επίσης, τέθηκε αυτό το ερώτημα πολλούς μήνες και δεν ασχοληθήκατε εδώ και μήνες. Θα ήθελα να μου δώσετε τώρα την απάντηση εκ μέρους της Επιτροπής. Διότι ίσως υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θα μπορούσαν να μου απαντήσουν. Αν κάποιος παρακολουθεί το όλο θέμα, το τώρα είναι θέμα αποφασιστικής σημασίας. Σήμερα στην ομάδα εργασίας μιλήσαμε για τους ε, ε, κινδύνους. Μιλήσαμε σήμερα το πρωί για κάποιους ε, θέματα που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε. 50% ε, ευθύνονται για τους καρκίνους, ευθύνεται το κάπνισμα τους καρκίνους. Δεν ξέρω αν αυτά είναι τα εξίσου υψηλά ποσοστά. Το να σταματήσει κανείς το κάπνισμα και να αρχίσει το ηλεκτρονικό τσιγάρο, μήπως μπορεί να εκλειφθεί κάποιος, κάποιος ως μια προτροπή να αρχίσουν ε, να, το άτμισμα. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε τα παιδιά και οι νέοι να μην αρχίσουν να καπνίζουν και να μην ε, βρουν ως εναλλακτική λύση αμέσως το άτμισμα. Θα ήθελα λοιπόν να μπορέσουμε γέρος να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Ξέρουμε ότι 50% των καρκίνων οφείλονται στο κάπνισμα, το επαναλαμβάνω. Θα ήθελα να ξέρω εάν πραγματικά το άτμισμα μειώνει αυτό το ποσοστό κινδύνου, διότι δεν έχουμε τέτοιου είδου στοιχεία, αλλά θέλω ενημέρωση. Διότι δεν θέλω να ενθαρρύνουμε άτομα να χρησιμοποιούν ένα προϊόν το οποίο εκ των υστέρων μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα υγείας. Στη ΣΥΠΑ τι ακριβώς γίνεται, μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς Σας ευχαριστώ. Ε, θα λάβω εγώ τώρα το λόγο εκ μέρους της Άντε. Στους τελευταίους μήνες έχουμε παραστεί σε μια κρίση η οποία πραγματικά προέρχεται από τη σμίσμα, ξέρουμε ότι έχουμε πέντε και παραπάνω ε, θανάτους στη ΣΥΠΑ, ένα στο Βέλγιο και προβλήματα. Από το 1,5% πέρασε στο σχεδόν 21% τελευταία χρόνια μεταξύ των νέων. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα δικά μας στην Ισπανία, η... τα νέα παιδιά 14 με 18 ετών ε, το 50 λοιπόν το έχουν ρίξει στο άπτισμα. Ο ΠΟΗ πολλές φορές μας είπε ποιες είναι οι επιπτώσεις της χρησιμοποίησης αυτών των προϊόντων και τα θεωρούν βλαβερά. Και πραγματικά ε, πρέπει να κάνουμε κάτι για να μειώσουμε και τη χρησιμοποίησή τους. Ε, είναι σαφές ότι κάτι τέτοιο δεν είναι κάτι το οποίο εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση το έχουμε λάβει ε, υπόψη. Σύμφωνα με τους ε, εμπειρογνώμενους είπαν ότι το... τα υγρά αναπλήρωσης, κάποια συγκεκριμένα, σίγουρα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Και βεβαίως ξέρουμε ότι υπάρχει κενό νομοθεσία για κάποια προϊόντα, δεδομένου ότι δεν έχουμε ολοκληρώσει προσπάθεια. Επίσης ένα έγγραφο εργασία για την οδηγία του 2011 για τις... Ε, ε, τη φορολόγηση για τον ε, καπνό Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Θα πρέπει να κάνουμε α, έρευνα και να μπορέσουμε σε όλα αυτά τα θέματα να συμπεριλάβουμε την ε, νόμιμη πώληση προϊόντων καπρού, τα, τα, την, ε, το ότι έχει σχέση με τα αυξημένα ποσοστά ε, καρκίνου, τα θέματα τα φορολογικά του παραεμπορίου και όλα τα σχετικά θέματα. Βεβαίω πρέπει να πω, όπω είπε και η Επιτροπή, ότι έχουμε διάφορε ελλείψει και θα ήθελα να ξέρω εάν προβλέπετε σε σχέση με το STBD ε, να κάνετε κάτι ώστε να μπορέσει αυτό το ε, κενό ε, που υπάρχει για τα υγρά αναπλήρωσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να το διορθώσετε. Παίρνω το λόγο εκ μέρους του συναδέλφου Φρέντερικ Ρίς, τη συναδέλφου, ε, η οποία είναι συγγήτρια για τα προϊόντα καπνού και που με παρακάλεσε να ε, θέσω κάποια ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα όμως ε, μία παρατήρηση για τα πιθανά τοξικά αποτελέσματα οποιοδήποτε προϊόντος. Όταν μιλάμε για τον καρκίνο, η χρονική περίοδος ε, στην οποία μπορεί να βρεθεί, να ανοιχνευτεί τοξικό αποτέλεσμα ενός προϊόντος είναι 10 χρόνια μετά την χρήση του. Ε, το θέμα λοιπόν είναι ότι θα ε, έπρεπε να έχουμε 10 χρόνια εμπειρία. Ε, έτσι είναι τα πράγματα δυστυχώς. Οι ερωτήσεις είναι οι εξής. Η Κομισιόν μπορεί να μας πει η Κομισιόν ότι δεν έχουν αναφερθεί παρόμοια περιστατικά σαν αυτά ε, με προβλήματα στους πνεύμονες των ΗΠΑ εκτός από την περίπτωση που αναφέρθηκε στο Βέλγιο. Ε, τώρα, ο κίνδυνος για τους μη καπνιστές που αρχίζουν να καπνίζουν ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ε, θα πάρει μέτρα η Κομισιόν ώστε να αποτρέψει την βιομηχανία από το να στοχεύει τους πιο νέους καταναλωτές. Η Κομισιόν θα λάβει υπόψη τις μελέτες, όπως αυτή από την Αγγλία, που δείχνουν ότι ε, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με αρώματα έχουν οδηγήσει σε ε, μείωση του καπνίσματος στους ενήλικες. Και επίσης η Κομισιόν στα πλαίσια της επανεξέτησης οδηγίας για τα προϊόντα καπνού το 2021 επιβεβαιώνει η Κομισιόν ότι θα διατηρήσει μια ισορροπημένη προσέγγιση, δηλαδή ότι θα αντιμετωπίζει το ηλεκτρονικό τσιγάρο σαν ένα μέσο σταματήματος του καπνίσματος και όχι σαν ε, μια εναλλακτική ως προς το παραδοσιακό κάπνισμα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Μπενέ. Μπενιού, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Δεν πειράζει. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η κατανάλωση καπνού μειώθηκε κατά 6% ανάμεσα στο 2006 και το 2017 σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Μια μελέτη στην έκθεση αντιξιών δείχνει ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι αποτελεσματικό τρόπος για να ε, σταματήσει κανεί με ήπιο τρόπο το παραδοσιακό κάπνισμα. Σύμφωνα με, μια, ε, σύμφωνα με την απαγόρευση του 2017, έχουμε απαγόρευση σε κάποιους δημόσιους χώρους και στο σχολικό περιβάλλον που κινούνται προς σωστή κατεύθυνση. Επιπλέον, όσον αφορά τα υγρά αναπληρώσεις, υπενθυμίζω στην Κομισιόν ότι κυκλοφορούν προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μη συμβατά προς την Ευρωπαϊκή ε, Νομοθεσία που οδηγούν σε τοξικά αποτελέσματα, σε δηλητηριάσεις. Υπάρχει ένα φάρμακο που ονομάζεται Μπουνταλού, το οποίο καταναλώνεται ε, στα ηλεκτρονικά ε, τσιγάρα, ε, πρόκειται για συνθετική κάναβη και δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα έκθεσης για την νεολαία. Τι κάνει λοιπόν η Κομισιόν ε, για τα προϊόντα που εισέρχονται παράνομα στον χώρο Σέγγεν και τι δράσεις θα αναλάβετε κατά της κυκλοφορίας του ναρκωτικού αυτού που ονομάζεται Μπουνταλού. Ευχαριστώ κυρία Μπένιε. Τώρα ε, δίνω το λόγο στην κυρία Ριλαζή για τους πράσινους. Ευχαριστώ. Όπως είπε προηγουμένως η Κομισιόν, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να κάνουμε τη διαφοροποίηση ανάμεσα στο ηλεκτρονικό τσιγάρο και στον θερμενόμενο ε, ή αεροποιημένο καπνό. Είναι διαφορετικά προϊόντα. Ο αεροποιημένος καπνός, αντίθετα με το ηλεκτρονικό τσιγάρο, περιλαμβάνει καπνό και άρα πρέπει να διαβέται από την ίδια νομοθεσία όπως τα παραδοσιακά τσιγάρα ή ε, τα στριφτά τσιγάρα. Επίσης πρέπει να δούμε και το θέμα της ε, φορολογίας των ηλεκτρονικών τσιγάρων, όπως γίνεται στην Λιθουανία. Ε, γίνεται με, πολλής λόγος για την μεταρρύθμιση της οδηγίας για τα καπνικά προϊόντα, αλλά πολύ λίγος λόγος για την ε, φορολογία των προϊόντων αυτών. Θα πρέπει η Κομισιόν να κάνει κάτι στον τομέα αυτό στο μέλλον. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι η σύνδεση ανάμεσα στο ηλεκτρο... η σχέση ανάμεσα στο ηλεκτρονικό τσιγάρο και την υγεία. Και θυμάμαι μια συζήτηση που έγινε το 2014 για την οδηγία για τα προϊόντα καπνού και εγώ ε, πέσα την προσοχή ενάντια στο γεγονό ότι αντιμετωπίζουμε σαν ένα μπανάλ, σαν ένα συνηθισμένο προϊόν το ηλεκτρονικό σιγάρο. Ενώ ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα για τα χημικά πρόσθετα που χρησιμοποιούνται, για το γεγονό ότι υπάρχουν κατάλοιπα ε, λόγω τη καύση που γίνεται εκεί, για τα συνδυασμένα αποτελέσματα, τα σωρευτικά αποτελέσματα. Ε, οι επαγγελματίε του κλάδου αναγνωρίζουν την άγνοιά του και θα ήθελα να ξέρουν περισσότερα πράγματα για τις πραγματικές συνέπειες των προϊόντων τους. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν γίνει η αναθεώρηση αυτής της οδηγίας θα πρέπει να πάρουμε πιο δρακόντια μέτρα και ε, να καταλάβουμε ότι δώσαμε άδεια στα προϊόντα αυτά με πολύ χαλαρό τρόπο. Ακούσαμε την Κομισιόν να λέει ότι περιμένει την επιστημονική γνωμοδότηση. Ναι, αλλά τι, πρέπει να την περιμένουμε όπως ένας ασθενής. Γιατί όταν βλέπουμε ε, τα νούμερα των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2.400 ασθενεί και κάποιοι ε, θάνατοι. Και έχουμε και ένα θάνατο στο Βέλγιο. Γιατί κάναμε αυτή την οδηγία για τον καπνό, για να μειωθεί η κατανάλωση ε, από τους νέους και βλέπουμε ότι δίνουμε ε, εγκρίσεις σε όσο δυνατόν πιο ελκυστικά αρώματα και γεύσεις για να προσελκύσουμε τους νέους στη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Απαγορεύουμε τα αρώματα για τον καπνό και επιτρέπουμε στα ηλεκτρονικά τσιγάρα να χρησιμοποιούν όσα αρώματα θέλουν. 25% λέμε... Ε, ε, των νέων χρησιμοποιούν το άτμισμα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, όταν κάποιο θέλει να σταματήσει το κάπνισμα, εγώ δέχομαι να ε, χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό ε, τσιγάρο για να απαλλαγεί από το κάπνισμα. Αλλά με του νέου το αποτέλεσμα είναι ακριβώ το αντίθετο και αυτό φυσικά ε, τους οδηγεί σε κέρδη ε, σε, στους, για τους παραγωγούς καπνού. Θέλουμε πιο δρακόντια μέτρα. Βλέπουμε οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν απαγορεύσει τη χρήση αρωμάτων. Η Κομισιό λοιπόν και αυτή πρέπει να απαγορεύσει τη χρήση των αρωμάτων. Αν ε, δεν θέλουμε να αποκτήσουν τη συνήθεια αυτή οι νέοι. Τώρα, ας δούμε στα κράτη-μέλη. Η Γαλλία είναι ο, η, ο δεύτερος χρήστης ηλεκτρονικού τσιγάρου μετά ε, τις Ηνωμένε Πολιτείε. Υπάρχουν δύο ουσίες που είναι προβληματικές στην ε, Γαλλία, ε, διασετίν και πέντα νοδιδιών, δύο-τρία. Η Γαλλία απαγόρευσε την πρώτη από αυτές τις ουσίες, γιατί διαπίστωσε ότι προκαλεί προβλήματα στους πνεύμονες, στον πνεύμονα, αλλά εσείς είπατε ότι αναθέσατε την αρμοδιότητα αυτή στα κράτη-μέλη. Η Γαλλία έχει την τύχη να έχει εμπειρογνώμονες ειδικού στα θέματα αυτά. Στα άλλα κράτη τι γίνεται. Ενθαρρύνεται η χρήση αυτών των ουσιών χωρίς να έχουν τα απαραίτητα μέσα να ελέγξουν τι ουσίες αυτές. Ε, ρωτάω λοιπόν την Κομισιόν. Τι μέτρα πιο δραστικά από αυτά που αναφέρατε θα πάρετε χωρίς να περιμένετε την αναθεώρηση τη οδηγία για το, τα προϊόντα καπνού. Πρέπει να απαγορεύσετε τη χρήση των αρωμάτων αν θέλετε να μην καπνίζουν οι νέοι πρέπει να γίνουν μελέτες για τα πρόσθετα και πάνω απ' όλα να χρησιμοποιηθεί η έρευνα, αλλά με το σωστό τρόπο. Γιατί είχαμε θανάτους στις ΗΠΑ, γιατί κάνουν μόνοι τους τι αναμίξει, τα μείγματα. Γίνεται εξατομικευμένη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Πρέπει να είναι πολύ πιο δραστικά τα μέτρα. Στη Γαλλία δεν ε, επιτρέπεται να γίνουν τέτοιε ε, ε, ε, ιδιωτικά. Άσε βέβαια που πολλά πράγματα περνάνε από το ίντερνετ. Ευχαριστώ. Ε, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, αλλά να μην μιλάμε και περισσότερο για από την Κομισιό. Εκ μέρου του ECR ο κύριο Φιόκ έχει το λόγο. Uh, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω. Είμαι μηχανικός. Θα ήθελα λοιπόν να έχω κάποια υλικά στοιχεία Έχω διαβάσει 24 διαφορετικές ακαδημαϊκές μελέτες για το θέμα του ατμίσματος, ε, σαν μια άλλη μορφή καπνίσματος και στην πραγματικότητα αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μπορεί κανείς εκεί να βρει τα πάντα και το αντίθετό τους. Ε, για να πάρω μια απόφαση πρέπει να έχω μια πραγματικά επιστημονική μελέτη σχετικά με το Πώς έχει αυτό το ζήτημα. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε το ηλεκτρικό τσιγάρο για να μειώσουμε το κάπνισμα ή αποτελεί ένα πραγματικό κίνδυνο για τους εφήβους που αρχίζουν με το άτμισμα και τελικά ε, έχουν προβλήματα με την υγεία τους. Θα ήθελα πραγματικά η Κομισιόν λοιπόν να ε, ξεκινήσει μια πραγματικά επιστημονική μελέτη για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφο. Κυρία Σαλτεμόσα. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στα αγγλικά γιατί δεν έχουμε δανέζικα σήμερα. Πρώτα απ' όλα ε, συνειδητοποιώ ότι μπορεί να είναι δύσκολο να πάρει μια απόφαση η Κομισιόν για το πώς να ενεργήσει τον τομέα αυτό λόγω της έλλειψης ε, ε, περιστατωμένων ε, επιστημονικών μελετών για τις συνέπειες. Όμως πρέπει να πω ότι πολλές από τις ε, αντικαρκυνικές εταιρείες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ζητούν πολύ πιο αυστηρά μέτρα κατά του ηλεκτρονικού τσιγάρου και του αεριοποιημένου καπνού. Αυτό δεν εντυπωσιάζει καθόλου την Κομισιόν ώστε να υιοθετήσει μια πιο αυστηρή στάση. Είπατε ότι δώσατε την αρμοδιότητα στα κράτη-μέλη να κάνουν τα σχετικά. Αλλά δεν θα ήταν καλύτερο και για ε, λόγους υγείας, αλλά και για λόγους της εσωτερικής αγοράς να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση και μια πιο αυστηρή προσέγγιση ε, και να μην βασιζόμαστε μόνο και να βασιζόμαστε στην αρχή της προφύλαξης περισσότερο σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και αργότερα αν έχουμε τις σχετικές ε, γνώσεις ε, και αποδείξεις θα μπορούσαμε να έχουμε μια πιο ανοιχτή στάση πάλι όταν αποδειχτεί ότι δεν υπάρχει ε, αρνητικός αντίκτυπος. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, δεν σας εντυπωσιάζει, δεν σας επηρεάζει το ότι οι αντικαρκυνικές εταιρείες όλη την Ευρώπη προτείνουν μια πιο αυστηρή στάση. Ευχαριστώ και πάλι εκ μέρους της Επιτροπής ο κύριος Ρης. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανησυχίες που ακούστηκαν. Πρώτα απ' όλα, ε, όταν βλέπετε τα στατιστικά στοιχεία, τα στατιστικά στοιχεία που δίνουμε ε, βασίζονται στο Ευρωβαρόμετρο του 2017 και στην ερώτηση που έγινε σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου από τους νέους. Τώρα βρισκόμαστε στην τελική φάση του Ευρωβαρομέτρου ε, του 2020. Ίσως ε, πειραματίστηκαν οι νέοι και με το τσιγάρο και με το ηλεκτρονικό τσιγάρο παράλληλα. Ίσως θα πρέπει να διευκρινίσουμε το σημείο αυτό για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτό το θέμα. Όπως ξέρουμε, η ιστορία αυτής της οδηγίας ε, ήταν ε, ότι η αρχική πρόταση της Κομισιόν ήταν πολύ πιο περιοριστική και πρότεινε ε, μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το ηλεκτρονικό τσιγάρο, αλλά τελικά καταλήξαμε στην οδηγία που έχουμε σήμερα ενισχύ, που είναι ένα μείγμα εναρμόνισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο με μέτρα παράλληλα που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη. Και νομίζω ότι η κρίση αυτή που προέκυψε στις ΗΠΑ οδήγησε ε, έναν αριθμό κρατών μελών να υιοθετήσουν ε, στάση πολύ πιο αυστηρή από ό,τι στο παρελθόν. Όπως αναφέρθηκε ήδη, βλέπουμε ήδη να γίνεται συζήτηση για την απαγόρευση των αρωματικών ουσιών ε, έχει γίνει ήδη αυτό σε ένα κράτο μέλο, θα δούμε και άλλα να, να ακολουθούν στους επόμενου μήνε. Επίσης υπάρχουν ενδιαφέρουσε ε, εξελίξει ε, και πρωτοβουλίες ε, με εκδηλώσεις που γίνονται στα σχολεία όπου εξηγούνται αυτά τα προϊόντα, τι συνέπειε μπορούν να έχουν και απευθύνονται και στα παιδιά και στους γονείς. Επίση, αναφέρθηκε το θέμα τη φορολογίας που είναι μια ενεξελίξη διαδικασία, μια συζήτηση. Όσον αφορά την έρευνα, προσπαθούμε πάρα πολύ, ξέρετε, η Επιστημονική Επιτροπή τι κάνει αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί να συλλέξει όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία και δεδομένα από όλε τι διαθέσιμε πηγέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από ερευνητέ, από τα κράτη-μέλη, μέσω τη συνεργασία μα ε, με το FTA, με, με συνεργασία με την Ιαπωνία. Προσπαθούμε να οικοδομήσουμε μία βάση αποδεικτικών στοιχείων. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι παρόλα υπάρχει ο ΠΟΗ, υπάρχει η FTCP που ε, ε, αναπτύσσουν παρόμοιες δραστηριότητες. Ελπίζουμε ότι στο κοντινό μέλλον θα έχουμε ε, μια ισορροπημένη ε, θέση σχετικά με το τι αποδίδει και τι δεν αποδίδει. Ε, μια ερώτηση που θέσαμε στην Υποστημονική Επιτροπή αφορά το σταμάτημα του καπνίσματος. Ε, είναι καλύτερο να προσπαθήσει κανείς να σταματήσει το κάπνισμα με τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Είναι μια υπόθεση που πρέπει να ελεγχθεί. Ε, υπάρχουν διάφορα άρθρα και μελέτες, αλλά δεν υπάρχουν ακόμα συγκεκριμένα συμπεράσματα στα οποία να βασίσουμε την θέση μας για το μέλλον και τις προτάσεις μας. Φυσικά, η Κομισιόν εφαρμόζει αυτά που αποφάσισαν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Έχουμε την ε, ε, οδηγία που είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Αυτό έχουμε μπροστά μας. Φυσικά εκτιμούμε και αξιολογούμε την κατάσταση στις Ηνωμένε Πολιτείες Σύμφωνα με μια μελέτη που έγινε στις Ηνωμένε Πολιτείε, στην αρχή τα πράγματα δεν ήταν πολύ σαφή, αλλά τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε πώς πρέπει να αξιολογηθούν αυτά τα περιστατικά, γιατί και όσον αφορά ε, την κλινική εικόνα, ήταν δύσκολο να συμφωνήσουν μεταξύ τους οι γιατροί για το πώς συνδεόντουσαν αυτά τα περιστατικά με το προϊόν. Τελικά όμως το συμπέρασμα είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα τα αποτελέσματα που προέκυψαν ε, με τα πνευμονολογικά προβλήματα ήταν αποτέλεσμα ενός συνδυασμού ε, της χρήσης δηλαδή και βιταμινών μέσα στο υγρό αναπλήρωσης και επίσης ε, της χρήσης κάναβης μες, ταυτόχρονα. Ε, αυτό λοιπόν ε, ε, α, επίσης υπήρχε ένα θέμα του μεγέθους των ε, δοχείων αναπλήρωσης που ήταν μεγαλύτερα από αυτά που επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε λοιπόν συνεχίζουν να καταβάλουν προσπάθειες για καλύτερη κατανόηση του φαινομένου. Στην Ευρώπη έχουμε και ένα σύστημα ειδοποιήσεων για να δούμε και το σύστημα που έχουμε για τον έλεγχο ε, των συσκευασιών στο RAPEX. Εκεί δεν υπήρχαν ε, ειδοποιήσεις. Ε, χρησιμοποιούμε και το σύστημα που έχουμε για τον έλεγχο ό,τι αφορά την υγεία του πληθυσμού και ούτε εκεί υπήρχε ειδοποίηση. Στο Βέλγιο βέβαια είχαμε την περίπτωση ασθενούς που χρησιμοποιούσε αυτό το προϊόν, όπως και στη ΣΥΠΑ. Είχαμε λοιπόν κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν επιβεβαιώθηκαν στην ε, κλινική εξολόγηση. Για να σας απαντήσω λοιπόν, δεν έχουμε αντίστοιχη κατάσταση στην Ευρώπη όπως έχουμε στις ΗΠΑ. Για πολλούς λόγους. Ποια είναι τώρα τα παραθυράκια στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τον κανονισμό ο καθένας με το δικό του τρόπο. Ταυτόχρονα όμως έχουμε τη δυνατότητα και να συναντιούνται, έχουμε ομάδες ε, με, όπου γίνεται μια ανταλλαγή απόψεων για τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού. Όχι μόνο για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, αλλά και για τον αεροποιημένο καπνό και, και για άλλα ζητήματα όπως η τοποθέτηση, ε, η διαφήμιση του καπνού, τα, ε, οι χώροι καθαροί από καπνό και το Και μεταξύ των υπήρων υπάρχει τέτοια συζήτηση για την ανταλλαγή απόψεων. Θέλουμε να δούμε πώς ε, και να ερευνήσουμε πώς κινείται η κατανάλωση καπνού και όλη αυτή η αγορά. Η βάση δεδομένων που θεσπίστηκε από αυτή την ε, οδηγία μας δείχνει ότι έχουμε 253.000 ε, ειδοποιήσεις προϊόντων. Δεν μιλούμε μόνο για ηλεκτρονικά τσιγάρα, αλλά και πολλά, πολλές άλλες συσκευές που παρασκευάζονται από διάφορες εταιρείε για αυτά τα προϊόντα. Είναι μια μεγάλη αγορά λοιπόν, με πολλές διαφορετικές μορφές. Πώς φτάνουν αυτά τα προϊόντα στην εσωτερική αγορά. Κάθε εταιρεία που τοποθετεί, που θέτει σε εμπορία ε, τα προϊόντα αυτά πρέπει να κοινοποιεί αυτή την πρόθεσή τη έξι μήνε εκ των προτέρων. Δεν υπάρχει δυνατότητα έναρξη των πωλήσεων χωρί αυτή την ειδοποίηση, χωρί αυτέ τι πληροφορίε. Υπάρχουν επιπλέον πληροφορίε στο προϊόν και μπορούν τα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν ε, το προϊόν αυτό ή να ζητήσουν επιπλέον πληροφορίε. Μπορούν να ζητήσουν πρόσθετα στοιχεία λοιπόν από την εταιρεία. για τις μελέτες που έχει κάνει η εταιρεία για το κάθε προϊόν. Αυτό είναι κάτι που ήδη γίνεται στις πολιτείες. Προς την κυρία Ριβαζή, ο αεριοποιημένο καπνό είναι προϊόν καπνού. Δεν είναι ηλεκτρονικό τσιγάρο. Είναι σημαντικό να το λέμε αυτό, γιατί συχνά με την ε, φορολογική ταξινόμηση και μετά από όλη αυτή τη συζήτηση αποφάσισαν τελικά να μπει αυτό το προϊόν στην ίδια κατηγορία με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Γι' αυτό θέσαμε αυτό το ερώτημα μέσω της FCTC και της COP για να κατανοήσουμε πραγματικά τι είναι αυτό το προϊόν. Θέλουμε την απάντηση της γραμματείας FCTC μέχρι το καλοκαίρι για να κατανοήσουμε καλύτερα το θέμα και να υπάρξει μια αναρμόνιση συνολικά. σε ό,τι έχει να κάνει με τον αεροπλανό καπνό και άλλα προϊόντα. Θα μπορούσε να είναι πιο περιοριστική η οδηγία. Κάποιες θέλουν να τα απαγορεύσουν, όπως στην Ινδία, ας πούμε. Αλλά είναι μια διαφορετική διαδικασία. Εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο στην νομοθεσία μας, πρέπει να σκεφτούμε και την αρχή της αναλογικότητας. Μπορούμε να κινηθούμε πιο γρήγορα με τα κρατημέλη από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς έχουμε το ρόλο του θεματοφύλακα, της νομοθεσίας, ε, την ανάληψη δράση σε περίπτωση που αυτό απαιτείται και την επικοινωνία με τα κρατημέλη. Αυτό κάνουμε θεωρούμε ότι τα κάτι μελη πλέον δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ανάληψη δράσης, ιδίω μετά τα όσα συνέβησαν στι ε, στις ΗΠΑ. Η τελική απόφαση όμως ε, θα βασιστεί στα δεδομένα που θα συλλέξουμε μέσα στους επόμενους μήνες. Όπως είπα και προηγουμένως, θα είμαστε σε θέση, θεωρώ, να αποστείλουμε έκθεση για την υλοποίηση της οδηγίας μέχρι την επόμενη άνοιξη και θα έχετε αρκετά στοιχεία για να συζητήσετε τι θα γίνει στο μέλλον. Ευχαριστώ. Muy bien, pues gracias, y a todos los... Καλά, ευχαριστώ τον κύριο Ρης και όλους τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο για το θέμα αυτό της ημέρης της διάταξης. Περνούμε τώρα στα επόμενα, 17 και 18. Έχουμε κοινή συζήτηση. Πρόκειται για δύο ειδικέ εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Πρώτα απ' όλα, για 10 λεπτά και εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το λόγο έχει ο κύριος Ζουάου Φιγκεραίδο. Thank you, Mr. Chairman. Um... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Περιβάλλοντος για την πρόσκληση που απίφθηνε στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για να σας ε, παρουσιάσουμε αυτή την ε, έκθεση ελέγχου για τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς, αλλά και για την έκθεση για, τα, ε, για τις εκπομπές του θερμοκηπίου που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Το πρώτο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να θίξω The first question I would like to raise... Το πρώτο ζήτημα λοιπόν που ήθελα να φέρω είναι γιατί προβήκαμε σε αυτό το εγχείρημα. γιατί πρόκειται για μια σημαντική πηγή πληροφοριών για τις περιβαλλοντικές πολιτικές, όπως ε, οι στόχοι για την βιώσιμη ανάπτυξη και το 7 σχέδιο περιβαλλοντικής δράσης. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι επικαιροποιημένες αξιόπιστε πληροφορίε είναι κέρια σημασία προκειμένου να παρακολουθούμε την ε, ε, πρόοδο προς την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Οι υπερβολητικοί λογαριασμοί είναι ένα στατιστικό πλαίσιο που περιγράφει τη σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και οικονομίας. Παράλληλα, η ποιότητα και συνάφεια των περιβαλλοντικών οικονομικών λογαριασμών είναι κρίσιμες σημασία για την μεγιστοποίηση του αντικτύπου τους. Γιατί λοιπόν αναλάβαμε αυτό τον έλεγχο, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν πολλά στάδια ε, σε αυτό το στατιστικό πλαίσιο καθώς και διάφορα εμπλεκόμενα μέρη σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλοι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν μέρους, ρόλους και αρμοδιότητες. Ένα άλλο ζήτημα που θα ήθελα να, θα ήθελα να θίξω έχει να κάνει με τα ερωτήματα που θέσαμε και τις απαντήσεις που λάβαμε σε αυτόν τον έλεγχο. Το βασικό ζήτημα, το βασικό ερώτημά μας ήταν εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε, διαχειρίστηκε και αξιοποίησε αυτό το στατιστικό πλαίσιο σωστά. Και για να λάβουμε την απάντηση ε, αξιολογήσαμε πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίστηκε την ανάπτυξη των ε, περιβαλλοντικών οικονομικών λογαριασμών και αν ε, πληρούν τις ανάγκες της ευρωπαϊκής στοχοθεσίας. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν στη συνέχεια τα βασικά μας ευρήματα. Πρώτο εύρημα παρατηρήσαμε ότι το στρατηγικό πλαίσιο των ε, περιβαλλοντικών οικονομικών λογαριασμών δεν είναι ακόμα αρκετά ολοκληρωμένο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ένα πλήρες ε, σύνολο δεδομένων που είναι απαραίτητα. Δεν υπάρχει έγγραφο ε, που θα αναφέρει τους, ε, τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες για την χάραξη πολιτικής και την παρακολούθηση. Είδαμε επίσης ότι οι ανάγκες ε, των περιβαλλοντικών λογαριασμών δεν διατυπώνονται σαφώς, καθώς δεν υπάρχουν και οι απαραίτητοι δείκτες για την χάραξη πολιτικής και παρακολούθηση. Μετά διαπιστώσαμε ότι η στρατηγική δεν συνοδεύεται από ένα συνολικό και ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Υπάρχει στρατηγική για τους οικονομικούς λογαριασμούς, αλλά... αλλά όχι ένα περιθετωμένο σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των στόχων. Και είδαμε ότι υπήρξαν ε, ε, στρατηγικές ε, που επαναλάμβαναν ε, τους στρατηγικούς στόχους για πάνω από μία δεκαετία. Δεύτερη κατηγορία ευρημάτων έχει να κάνει με τις ανεπάρκειες που εντοπίσαμε. τέτοιες ανεπάρκειες και, και ελλείψεις ε, που αφορούσαν ε, τους περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς ε, και μείωναν έτσι την συνάφειά τους για την χάραξη πολιτικής. Η Επιτροπή λοιπόν δεν είχε μία πλήρη ανάλυση κόστους ωφέλους. Και είδαμε ότι η εφαρμογή του σχετικού πλαισίου πήρε πάνω από 10 χρόνια δεν αξιοποίησε αυτά τα πλαίσια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλες τις ε, πολιτικές, σε όλους τους συναφείς τομείς πολιτικής. Είδαμε ότι τα προγράμματα αυτά, τα πλαίσια αυτά δεν αξιοποιήθηκαν στο έπακρο για την παρακολούθηση βασικών πολιτικών όπως είναι η βιώσιμη στοχή ανάπτυξης και το 7ο σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και ορισμένα τέτοια προγράμματα δημοσιοποιήθηκαν ξεχωριστά και έτσι δεν μπορούσε κανείς να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Οι βασικοί χρήστες χρησιμοποιούν διαφορετικά σύνολα δεδομένων. Τέλος, υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία. Πρέπει να δούμε λοιπόν ότι η Eurostat αντιμετωπίζει προκλήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την συλλογή επίκαιρων και υψηλής ποιότητας δεδομένων. κάποια συλλογή δεδομένων γινόταν πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε. Δεν αξιοποιήθηκαν όλες τις δυνατότητες για την συλλογή επίκαιρων ε, στοιχείων. Δεν υπήρχε ε, χρονοδιάγραμμα για να γνωρίζουν οι χρήστες ε, πότε θα είναι διαθέσιμα τα δεδομένα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα των δεδομένων, δεν υπήρχαν επαρκείς πληροφορίες ε, που θα βοηθούσαν τη Eurostat να αξιολογήσει σωστά την ποιότητα των δεδομένων. Και είδαμε ότι η Eurostat ε, ε, επέλυε προβλήματα που ήγηραν τα κράτη-μέλη, αλλά δεν υπήρχε καθοδήγηση για μεθοδολογικά προβλήματα. Είναι κάτι το οποίο έπαιρνε πολλά χρόνια και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα δεδομένων. Βάσει αυτών των ευρημάτων καταλήξαμε σε ορισμένες συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει να κάνει ακριβώς με αυτές τις ε, αδυναμίε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να βελτιώσει το στρατηγικό πλαίσιο για τα δεδομένα που ε, συλλέγονται για τους περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς. Θα πρέπει επίσης η Επιτροπή να βελτιώσει την συνάφεια των ε, πλαισίων για, αυτά για αυτούς τους λογαριασμούς για τη χάραξη πολιτική, καθώς και, την το επίκαιρο αυτό των στοιχείων που συλλέγονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε τις συστάσεις μας και φαίνεται ότι έχουν αρχίσει ήδη να τις υλοποιούν, το οποίο είναι πολύ θετικό. Να επισημάνω επίσης ότι η συνεργασία του ελεγκτικού συνεδρίου με την DGNV και με την Eurostat ήταν εξαιρετική και μας βοήθησε να ολοκληρώσουμε αυτό το ελεγκτικό μας έργο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Φεγγερέδη για την δεύτερη έκθεση. Ο κύριο ε, Γενικός Διευθυντής, κύριος Πίτερ Βουέλκ. Ευχαριστώ. Χάνετε το μικρόφωνο το μιλητή. Um, uh, yes, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεδομένων των αρμοδιοτήτων του πρώτου τμήματο του Ελληνικού Συνεδρίου, ε, είναι σημαντική ευκαιρία για μα να ερχόμαστε εδώ και να μιλούμε για αυτά τα ζητήματα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη βιώσιμη χρήση των ε, φυσικών πόρων, τα θέματα του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, ε, είναι ζητήματα τα οποία μας ενδιαφέρουν ε, ιδιαίτερα. Σήμερα θα σας μιλήσω για μία έκθεση που δημοσιεύσαμε το Νοέμβριο του 2019 Αριστερά στο γράφημα βλέπετε το σημαντικό σκέλος, την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα. Να σας θυμίσω ότι όταν μιλούμε για εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, σαφώς και μας ε, αποσχολεί ιδιαίτερα το διοξίδιο του άνθρακα, αλλά έχουμε και εκπομπές μεθανίου, που είναι πολύ σημαντικές και είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια αυτής της έκθεσης. Εδώ βλέπετε ένα γράφημα ε, που παρουσιάζει την πρόοδο που έχει γίνει μέχρι τώρα, που είναι σημαντική και θεωρούμε ότι θα πετύχουμε το στόχο του 20% μείωσης ε, μέχρι το τέλος χρονιάς και βέβαια υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις για το μέλλον. Θα απαιτηθούν πολύ υψηλότερες προσπάθειες. Έχουμε μια έκθεση διασφάλισης ποιότητας στην ουσία. Βλέπουμε δηλαδή τι γίνεται στα κράτη-μέλη για την συλλογή αξιόπιστων στατιστικών ε, στοιχείων. Επικεντρωνόμαστε στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μαζί και με τον ε, Οργανισμό Περιβάλλοντος στην Κοπεχάγη Όλα αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας, αλλά εμείς βασιζόμαστε σε στοιχεία που έχουν συλλεγεί από έξι κρατημέλη, Γερμανία, Τσεχία, Ιταλία, Γαλλία, Πολωνία, Ρουμανία. Και έχουμε καταγράψει και το έργο της UNFCCC. Περνώ στα ευρήματα. Ξεκινώ από τα θετικά. Είδαμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σωστά ελέγχει και υποβάλλει εκθέσεις ε, για τα δεδομένα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά τις εκπομπέ, σύμφωνα και με το πρωτόκολλο του Κιώτου και τι κατευθύνες γραμμέ IPCC. Ακόμα και πέραν ε, των ε, απαραίτητων, παρέχει στοιχεία για τον αντίκτυπο της αεροπλοείας πέραν του διοξιδίου του άνθρακα, για παράδειγμα, και στο φορά το αποτύπωμα άνθρακα. Η ποιότητα των δεδομένων βελτιώνεται έχουμε λιγότερες διορθώσεις και βλέπουμε ότι και τα κράτη-μέλη ε, εκτιμούν τις ε, κατευθύνσεις αυτές που τους δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά είναι τα θετικά. Τώρα, υπάρχουν και άλλοι τομείς βέβαια, όπου απαιτείται μεγαλύτερη ε, πρόοδο. Σίγουρα ένα από τα λιγότερο θετικά σκέλη είναι το ΛΟΥΛΟΥΣΙΕΦ, η χρήση γης, αλλαγή στη χρήση τη γης και τι οικονομικέ δραστηριότητε. Μέχρι το 2030 εντάσσεται στον ε, στόχο, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε μέχρι τώρα. Θέλουμε λοιπόν αυτό ο τομέας πολιτικής ΛΟΥΛΟΥΣΙΕΦ, να, ε, να τύχει τη ίδια αντιμετώπιση, όπω άλλοι τομεί ε, πολιτική για να πετύχουμε τον στόχο μέχρι το 2030. Υπάρχει αρκετά μεγάλη αβεβαιότητα σε αυτόν τον τομέα που είναι κρίσιμο σημείο για το μέλλον. Γιατί μακροπρόθεσμα θεωρώ ότι ο στόχος ε, και η επίτευξή του θα εξαρτηθεί και από την επιτυχία στη, στον τομέα Λουσέφ. Πρόκειται για μια καλή ευκαιρία περαιτέρω προόδου με τη χρήση των, της τεχνολογίας, με την παρακολούθηση μεσοδορυφόρου, Ας προχωρήσουμε τώρα. Πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη οπτική για το, για το μέλλον. Είναι θετικό που έχουμε ευρωπαϊκούς στόχους που καλύπτουν όλους τους κλάδους και όλα τα αέρια εκτός από το Λουλουσιεφ και εκτός από την διεθνή ναυτιλία. Είναι κάτι το οποίο συζητήσατε προηγουμένως. Υπάρχουν οδικοί χάρτε σε πολλού βασικού τομεί, αλλά είδαμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο οδικό χάρτη για τη γεωργία ή για τον Λουλουσιεφ. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ε, κέρια σημασία στοιχείο. Στο πλαίσιο υποβολή εκθέσεων, τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παράσχουν εκτιμήσεις για τον αντίκτυπο των ε, μέτρων που προτείνουν και υιοθετούν. Έχουμε εκ των προτέρων εκτιμήσεις από την Ευρωπαϊκή Τροπή για την πλειοψηφία των ε, κλιματικών ε, μέτρων, περίπου στα δύο τρίτα. Υπάρχουν και εκ των υστέρων δείκτες για τα δύο πέμπτα των πολιτικών και μέτρων που υιοθετούνται. Όμως, βλέπουμε ότι δεν έχουμε εκτιμήσεις για τον αντίκτυπο ορισμένων βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως είναι το σύστημα ανταλλαγή εκπομπών, το ETS, και ο αγροτικός ε, τομέας, η κοινή γεωργική πολιτική. Πολύ λογικά λοιπόν καταλήγουμε σε ορισμένες συστάσεις, όπως είναι η ενίσχυση των ελέγχων για τον τομέα Λουλουσιεύ και η ευθυγράμμιση με τους άλλους τομείς. Θέλουμε η Επιτροπή να θίξει και το ζήτημα της διεθνούς ναυτιλίας. Θεωρούμε πολύ σημαντικό τα στρατηγικά σχέδια για την Γεωργία και το LULUCF να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων μείωσης εκπομπών μέχρι το 2050 και θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει και να υποβάλει εκθέσεις προς την UNFCCC σε ό,τι έχει να κάνει με τον αντίκτυπο των εκπομπών σε όλους τους βασικούς τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή υπάρχουν και πολλές αλληλεπεκαλύψεις, δεν γίνεται να υπάρχει τέτοια έκθεση για όλους τους επιμέρους τομείς πολιτικής, αλλά για τους βασικούς τουλάχιστον. Κλείνοντας λοιπόν, τα θετικά είναι ότι έχουμε ε, ανταπόκριση σε ό,τι έχει να κάνει με τα διεθνή πρότυπα και βελτιωνόμαστε. Θα πρέπει όλα αυτά να ολοκληρωθούν βέβαια στο μέλλον, γιατί χρειάζεται αναβάθμιση των προσπαθειών μας σε ό,τι έχει να κάνει με τα όσα δεσμευόμαστε και με τα όσα πραγματοποιούμε. Και πρέπει να εξετάσουμε ε, και τον αντίκτυπο των εκπομπών σε άλλες ε, βασικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Συνάδελφοι που ζητούν το λόγο. Η κυρία Σπουδέτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τα αέρια θερμοκοινού είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που μας απασχολήσουν σήμερα. Η Επιτροπή ανέπτυξε, όπως είπατε, διάφορους χάρτες οδικής πορείας ώστε να μπορέσουμε να ασχοληθούμε τη μείωση των εκπομπών. Αλλά δεν υπάρχει κάτι το ειδικό για τον τομέα της γεωργίας, γιατί σύμφωνα με την ΦΑΟ, διότι η βιομηχανική γεωργία παράγει το 40% του ποσοστού εκπομπής θερμοκηπίου πράγμα, το οποίο αντιστοιχεί με αυτό που δημιουργείται από τον τομέα των μεταφορών. Προσπαθεί να κάνει μια πάρα πολύ φιλόδοξη Green Deal πολιτική η πολιτική, όπως η Επιτροπή. Όπως όμως λέγεται, δεδομένου ότι η, γεωργική πολιτική δεν μας δίνει δυνατότητες να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε τα θέματα των εκπομπών, πώς μπορείτε εσείς να ενεργήσετε ότι να ρυθμιστεί αυτό το θέμα εκ μέρους του Ελεκτικού Συνεδρίου. Η κυρία ο Σάλιβαν εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Το ερώτημά μου είναι όσον την ε, μέτρηση. Ξέρουμε ότι το ποσοστό ανθεκτικότητας είναι κάτι το οποίο κυρίως για την θάλασσα και για τους ωκεανούς είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι μπορεί να απορροφήσει ένα μεγάλο ποσοστό και μπορεί να δεσμεύσει κάθε χρόνο μεγάλα ποσοστά των ετησίων εκπομπών. Πιστεύετε ότι το οικοσύστημα blue carbon όπως λέγεται είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει, είναι θέμα για το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε μία σαφή εικόνα. Ποιες είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να ε, ενεργήσουν ώστε να προστατεύουμε ε, από την κλιματική αλλαγή και από τα προβλήματα που υπάρχουν τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του Έλκη, κυρία Νόβακ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πάρα πολύ πλήρη παρουσίαση που έγινε εκ μέρους ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε πάρα πολύ καλές στατιστικές για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε τα μέτρα που θα λάβουμε και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο αν ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα ώστε να εξεύρουν τις κατάλληλες Επίση, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τα μέτρα τα οποία προτείνετε λάβει η Επιτροπή σας συγχαίρω. Διερωτώ με όμως αυτές τις συστάσεις τις οποίες εσείς αποστήλατε αντέδρασε η Κομισιό ή έδωσε κάποια συνέχεια. Πώς ανταποκρίθηκε σε αυτές. Επίσης, θα ήθελα να μας στείλετε τα πιο αξιόπιστα στοιχεία που, διαθέτεται, διότι, που διαθέτετε, διότι πολλές φορές έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη οι πολίτες μας στη πορίσματα διεθνών μερετών παρά εθνικών. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι αξιόπιστα όλα αυτά τα στοιχεία και να τα έχουμε στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που έκαναν τις ερωτήσεις αυτές. Θα ήθελα ο Πίτερ Βέλς να απαντήσει την ερώτηση που αφορά τις εκπομπές καυσαρίων θερμοκηπίου και τα θέματα της ποικιλότητα. Ξέρω ότι έχουμε κάποιο χρόνο, μπορεί όμως να σας δώσει κάποια στοιχεία πιο συγκεκριμένα. Εγώ θα ήθελα τώρα να απαντήσω στο ερώτημα που τέθηκε για τις στατιστικές. Και με ποιο τρόπο και πότε η Επιτροπή θα προετοιμαστεί για τις νέες αλλαγές, ώστε να ανταποκριθεί και να απαντήσει στις συστάσεις που αποστήλαμε. Όπως είπα στην πρώτη μου παρέμβαση, η Επιτροπή δέχτηκε όλες τις συστάσεις που αποστήλαμε και μας έδωσε κάποιες πληροφορίες για την εφαρμογή τους. Μπορώ λοιπόν να πω ότι στον τομέα αυτό Υπάρχει χώρος για λήψη υποφάσεων. Υπάρχει μία συνεδρίαση που λέγεται τη Μέζα, στην οποία ε, συνεδριάζουν σε εθνικό επίπεδο υπεύθυνοι των στατιστικών υπηρεσιών και φέτος στην εν λόγω συνεδρίαση μελετήθηκε το όλο θέμα των συστάσεων και έχουν αρχίσει οι υπεύθυνοι να κάνουν κάποιες αλλαγές ώστε να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν. Οι συστάσεις λοιπόν αυτές πρέπει να πω ότι δεν έγιναν αποδεκτές μόνο από τη Eurostat και από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, αλλά διαβιβάστηκαν στους υπεύθυνε αρχές στατιστικών υπηρεσιών, οι οποίοι τις μελετούν και τις επεξεργάζονται. Όσον αφορά το θέμα των εκπομπών θα ήθελα να απαντήσει ο συνάδελφος. Ευχαριστώ. Πρώτη ερώτηση την οποία θα απαντήσω είναι τι θα κάνουμε στο μέλλον όσον αφορά την όλη εποπτεία και μελέτη που θέλουμε να κάνουμε στον τομέα τη γεωργία, κυρίω όσον αφορά το θέμα αυτό. Δεν θέλω να υπόσχεμαι πράγματα τα οποία θα κάνουμε, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε κάτι για την αντίκτυπο τη βιοπικιλότητα ε, τους επόμενους μήνες. Τέθηκαν πάρα πολλά θέματα ε, για την γεωργία και για τις εκπομπές θερμοκηπίου και νομίζω ότι το παρακολουθούμε το θέμα αυτό διότι μας ζήτησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εξετάσουμε τι γίνεται στον τομέα αυτό. αυτό συνδέεται με θέματα και βεβαίως ε, όταν θα έχουμε τις απαντήσεις εκ μέρους της Επιτροπής θα περάσουμε και θα σας ενημερώσουμε. Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει μέσα στο επόμενο εξάμεινο και θα παρακολουθήσουμε το του σήμα τι γίνεται. Τώρα, όσον αφορά τους ωκεανούς που αναφέρει συνάδελφό σας, είναι τρομακτικό το όλο θέμα. Τι Υπάρχει δηλαδή στο βάθος των ωκεανών, τι απορροφούν οι θάλασσες. Αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί όλους. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το μελετήσουμε το θέμα, να δούμε τι ακριβώς γίνεται στις παράκτιες περιοχές. Ε, ξέρουμε ότι οι τρομερές πλημμύρες που συνέβησαν τους τελευταίους μήνες επίσης πρέπει να μας κινητοποιήσουν το εξετάζουμε. Όσον αφορά την ανταπόκριση της Κομισιόν στις, συστάσεις μα μας για το αν βελτιώνουν τα πράγματα, νομίζω ότι στις εκθέσεις μας είπαμε ότι υπάρχει πολύ καλή ανταπόκριση εκ μέρους της Επιτροπής, διότι ακολουθεί τις συστάσεις μας πολλές φορές σε άλλες περιπτώσεις δεν θέλησε να ακολουθήσει τις συστάσεις μας, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα μας ακολουθεί. Άρα ό,τι κάνουμε νομίζω ότι συνεισφέρει στο να έχουμε μια συνενετική και κοινή στάση σε σχέση με το θέμα αυτό και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Ολοκληρώθηκε τώρα και η συζήτηση για αυτό το θέμα. Και περνούμε στο 19, στο τελευταίο τη σημερινή μερική διάταξη. Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με τα βλήματα που περιέχουν μόλιβδο. Το λόγο εκ μέρου τη Κομισιόν το έχει ο υπεύθυνο διευθυντή τεχνολογία, ο κύριο Πετινέλη. Yes, uh, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που καλέσατε την Κομισιόν για την ανταλλαγή αυτή απόψεων και που μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τη συνεχιζόμενη εργασία μας για το θέμα των βλημάτων με μόλιβδο. Έχω αυτές τις ε, διαφάνειες εδώ γιατί είναι αρκετά τεχνικό το θέμα. Λοιπόν, πριν ε, σας παρουσιάσω σε ε, την εργασία αυτή που εξελίσσεται στα πλαίσια του κανονισμού REACH, θα ήθελα να σας εξηγήσω κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που θα σας επιτρέψουν να καταλάβετε καλύτερα το θέμα. Λοιπόν, ο ορισμός. Γιατί πράγμα μιλάμε. Ένα ε, shotgun είναι ένα δίκανο το οποίο χρησιμοποιείται με μία μοναδική βολή που αδειάζει την κάνει. Χρησιμοποιείται κυρίως για κυνήγι και αριστερά μπορείτε να το δείτε στη διαφάνεια. Και πώς είναι το βλήμα του, το shot στα αγγλικά. Δεξιά στην ε, διαφάνεια είναι μια καραμπίνα. Η καραμπίνα ε, είναι ένα ε, όπλο που χρησιμοποιεί σφαίρες που είναι συμπαγή βλήματα. Άρα, συνολικά, για όλα αυτά, ε, όρος που χρησιμοποιείται στα αγγλικά είναι ammunition. Πολεμοφόδια. Τώρα, γιατί θέλουμε να περιορίσουμε την ε, ελευθέρωση μολύβδου στο περιβάλλον. Όπως ξέρετε, ο μολύβδος είναι μια ουσία πάρα πολύ τοξική για τους ανθρώπους και για την ε, ζωή γενικά. Εκτιμούμε ότι μεταξύ 18 και 20.000 τόνοι μολύβδου απελευθερώνονται κάθε χρόνο στο περιβάλλον από το κυνήγι που γίνεται με χρήση τέτοιων βλημάτων που περιέχουν μόλυβδο. Αυτά που βλέπουμε δηλαδή στην αριστερή μεριά της διαφάνειας. 4 με 5.000 τόνοι από αυτούς είναι, ε, απελευθερώνονται σε υγροβιότοπους και εκτιμάται ότι η δηλητηρίαση από μόλιδο σκοτώνει ένα εκατομμύριο πτηνών κάθε χρόνο στους υγρότοπους και με μια προκαταρτική εκτίμηση και άλλα πολλά εκατομμύρια πουλών έξω από τους υγροβιότοπους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και, τα 23 κράτη, και 23 κράτη μέλη της είναι μέλη της ε, σύμβασης ADWA με την Αφρική για την προστασία των μεταναστευτικών ειδών ε, που ε, περιλαμβάνει απαγόρευση της χρήσης των πλημάτων με μόλυβδο στους υγροβιότοπους το γρηγορότερο δυνατό ε, ένα αριθμό κρατών μελών ήδη έχουν νομοθεσία ε, για τον περιορισμό των πλημάτων αυτών, αλλά όχι με συνεκτικό τρόπο μεταξύ του. Αυτό λοιπόν ε, σημαίνει ότι απαιτείται ένα διαφορετικό, ότι υπάρχει διαφορετικό επίπεδο προστασίας. Όμως τα μεταναστευτικά είδη δεν μπορούν να επιλέξουν τους υγροβιότοπους όπου δεν υπάρχει μόλυβδος ή πολύ λίγος μόλυβδος. Αυτό απαιτεί λοιπόν μια εναρμόνιση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα υγεία των πτηνών και ε, ο άνθρωπος μπορεί να εκτεθεί στον μάλιβδο, στο μόλιβδο που προκύπτει από την κυνηγητική δραστηριότητα και ε, κατά την ίδια τη δραστηριότητα αλλά και από την διάχυση του μολύβδου στο περιβάλλον. στα πλαίσια του ΡΙΣ, λοιπόν, υπάρχουν δύο διαδικασίες περιορισμού του χρήση του μολύβδου. Ε, η πρώτη διαδικασία περιορίζει τη χρήση των βλημάτων ε, που βλέπουμε αριστερά, που περιέχουν μολύβδο, δηλαδή, ε, μόνο στους υγροβιότοπους. Η εργασία αυτή έχει προχωρήσει αρκετά καλά όσον αφορά αυτόν τον περιορισμό, στα κινητικά όπλα δηλαδή. Ο δεύτερος περιορισμός αφορά τη χρήση και εμπορία σε άλλες περιοχές εκτός των υγροτόπων ή άλλων είδων ε, πολεμοφοδίων που περιλαμβάνουν μόλιβδό, ε, όπως μέσα στις σφαίρες που βλέπουμε στα δεξιά στη διαφάνεια και τελικά ε, μιλάμε και για είδη ψαρικής που ε, χρησιμοποιούνται στο υγρό περιβάλλον, άγιστρα, βαρύδια και τεχνητά δολώματα που ε, παρουσιάζουν τον ίδιο κίνδυνο. Σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, η ε, Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό που ασχολείται με τα χημικά προϊόντα να ε, ορίσει τέτοιους περιορισμούς. Σας μιλάω τώρα για την ε, διαδικασία που ακολουθείτε. Λοιπόν, Ποια είναι η διαδικασία. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει ε, την, ε, από την ΕΚΑ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Ουσιών, να ε, ετοιμάσει μία γνωμοδότηση. Έχει χρόνο για να κάνει την εργασία αυτή η ΕΚΑ 12 μήνες μετά την υποβολή του αιτήματος. Η ΕΚΑ είναι έχει, έχει δύο επιστημονικέ επιτροπές, την Επιτροπή αξιολόγηση του Κινδύνου και την Επιτροπή Ανάλυσης ε, των Κοινωνικο-Οικονομικών Επιπτώσεων. Περιλαμβάνει εκεί, ε, περιλαμβάνουν οι επιτροπές αυτές ε, ε που έχουν οριστεί από τα κράτη-μέλη που πραγματοποιούν αντίστοιχα την ανάλυση κινδύνου και την κοινωνικο-οικονομική ανάλυση. Έχουν ε, 12 με 14 μήνες για την έκδοση αυτών των γνωμοδοτήσεων, όπως βλέπετε εδώ στη δεύτερη ε, γραμμή του πίνακα αυτού. Ε, η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει δημόσια διαβούλευση, όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα, σχόλιά τους. Η δημόσια διαβούλευση λαμβάνει η χώρα πριν οριστικοποιηθούν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Μετά από όλα αυτά τα βήματα, οι τελικές ε, επιστημονικές γνωμοδοτήσεις υποβάλλονται στην Κομισιόν. Αν αποδειχθεί ότι υπάρχει ένας αποδεκτός κίνδυνος για τον άνθρωπο ή για το περιβάλλον, μη αποδείκτο συγγνώμη κίνδυνος ε, για το περιβάλλον για τον άνθρωπο, η Κομισιόν ετοιμάζει μία πρόταση ε, περιορισμού της χρήσης. Στην επόμενη γραμμή εδώ. Βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση τώρα της προτινόμενης απαγόρευσης για την ε, κυνηγετική χρήση ε, μόνο και μόνο σε υγρότοπους. Η διαδικασία έχει προχωρήσει αρκετά και έχει καταρτήσει ήδη, έχει ετοιμάσει η Κομισιόν την πρόταση περιορισμού και τη συζητάει με τα κράτη-μέλη στην Επιτροπή ΡΙΤΣ. Βρισκόμαστε στην τέταρτη αράδα αυτής της διαφάνειας ενημερώνεται συνεχώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις αυτές μέσω του, της, επιτροπής, ε, επιτροπο, της διαδικασίας επιτροπολογίας. Μέχρι στιγμής ε, συνεχίζονται οι συζητήσεις με τα κράτη-μέλη και δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αρκετό βαθμό συνένεσης για να έχουμε μια επιτυχή ψηφοφορία στην Επιτροπή ΡΙΤΣ. Τα κύρια θέματα προς συζήτηση είναι τα ίδια με αυτά που έχετε θέσει εσείς σε διάφορες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Δηλαδή, ποιος είναι ο ορισμός του υγρότοπου, ποιο, ποιο, ποιο είναι το μέγεθος της ζώνης ανάσχεσης γύρω από, τις, από τους υγρό, υγρότοπους και ποιος πρέπει να ε, υπόκειται σε αυτούς τους κανόνες. Βρισκόμαστε στην πέμπτη γραμμή αυτής της διαφάνειας. Λοιπόν, περιμένουμε τα κράτη-μέλη στην Επιτροπή Ρίτζ να ψηφίσουν μια τελική πρόταση ε, κατά τους επόμενους μήνες. Ε, έχουμε τη διαδικασία την κανονιστική με έλεγχο. Δηλαδή, αν είναι θετική η ψηφοφορία αυτή, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχουν μια περίοδο τριών μηνών για να ελέγξουν τα μέτρα αυτά. Αν Κάποιο από του δύο έχει αντίρρηση, η Κομισιόν δεν μπορεί να υιοθετήσει αυτά τα μέτρα. Αυτό έγινε ήδη την περασμένη εβδομάδα όταν το Κοινοβούλιο αντιτάχθηκε ε, σε μία ε, πρόταση τη Κομισιόν για τον υπολοιπόμενο ε, μόλιβδο. Αυτό είναι ο πρώτο περιορισμό. Ο δεύτερο περιορισμό που θέλουμε να επιβάλλουμε για τη χρήση του μολύβδου εκτό των υγροτόπων και για άλλα είδη πολεμοφοδίων όπω είναι οι σφαίρε για άλλα όπλα και ε, για τα είδη ψαρικής. Βρισκόμαστε σε πολύ αρχικό στάδιο. Ζητήθηκε τον Ιούλιο του 19 από την Κομισιόν να ετοιμάσει ε, τη σχετική πρόταση. Μετά από μια έκθεση του Σεπτεμβρίου του 18 που έδειχνε ότι υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις για να ε, προταθούν περιοριστικά μέτρα και στις περιπτώσεις αυτές για χρήση τέτοιων όπλων στην ξηρά. Ε, αναμένεται ε, το ντοσιέ να ε, το έχουμε φέτος το Οκτώβριο. θα ξεκινήσει την εργασία της η ΑΕΚΑ, η Επιστημονική Επιτροπή, με, ξεκινώντας με τη δημόσια διαβούλευση όλων των ενδιαφερομένων μερών και αρχές του 2021 ή μάλλον προς τα τέλη του 2021 ή αρχές του 2022 θα φτάσει η σχετική γνωμοδότηση στην Κομισιόν. Άρα ε, για τη δεύτερη αυτή απόφαση ε, περιορισμού βρισκόμαστε στην πρώτη ε, σειρά αυτής της διαφάνειας, στην αρχική φάση. Σταματώ εδώ και είμαι ανοιχτό για να απαντήσω στις ερωτήσεις, στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πετινέλη. Ο κύριος Λίζε πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ, πολύ. Ευχαριστούμε για τον εκπρόσωπο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρώτη περίπτωση είναι αρκετά απλή. Υπάρχει μια διεθνής ε, σύμβαση. 24 κράτη-μέλη την εφαρμόζουν. Και είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξει αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας στους ε, υγροβιοτόπου. γιατί ο μόλυβδο έχει πολύ σοβαρέ επιπτώσει στο περιβάλλον. Και χαίρομαι που έχουμε χρόνο για τα άλλα μέτρα, γιατί πρέπει να διατηρήσουμε μια στάση αναμονής, να δούμε τον ε, περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καθώ και τι επιπτώσει για την υγεία. Εάν δεν υπάρχουν επιπτώσει, γιατί όλα αυτά συμβαίνουν εντός ενός προστατευόμενου περιβάλλοντος. Δεν πρέπει να ε, υιοθετήσουμε υπερβολικά αυστηρά μέτρα. Πρέπει να βρούμε ακριβώς που έχουμε ε, ε, συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία και να τα αντιμετωπίσουμε. Αλλά η πλήρης απαγόρευση του μολύβδου σε κάθε είδους πυρομαχικού και κυνηγετικού όπλου θα ήταν υπερβολική. Γι' αυτό θα απευθύνω μια έκκληση προς την Επιτροπή να καταλήξει σε μια ισορροπημένη πρόταση και να επικεντρωθεί σε τομείς όπου υπάρχουν πιθανές συνέπειες ε, για το περιβάλλον και την υγεία. Κύριε Μαγκίνες έχει τον λόγο. Ευχαριστώ. Ελπίζω να έχω λίγο χρόνο, γιατί υπάρχουν ε, πολλά ζητήματα που έχουν, ε, έχει θίξει ο Σύλλογος Κυνηγών στην Ιρλανδία. ευχαριστώ τους συναδέλφους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση και τη συνεργασία με το επιτελείο μου για αυτό το θέμα. Τα τρία στοιχεία που εντοπίσατε για τον ορισμό των υγροβιοτόπων, ε, το μέγεθος των ζωνών ενάσχεσης και των χρονομετάβασης, ε, όπου εκεί δυσκολεύεστε να βρείτε επαρκή ε, στήριξη στην Επιτροπή. Θα ήθελα να μου δώσετε περισσότερα στοιχεία, γιατί ο ορισμός του υγροβιοτόπου σίγουρα είναι θέμα προβληματισμού για πολλούς κυνηγού στην Ιρλανδία για το είδος εδαφών που καλύπτονται, όπως είναι τα οι τυρφώνες, οι στεγνοί τυρφώνες. Μετά, υπάρχουν στεναρές αντιστάσεις προς αυτή την υποτιθέμενη πλήρη απαγόρευση των ε, βλημάτων ε, και σφαιρών μολύβδου. Λένε ότι δεν λαμβάνεται υπόψη ε, το συμφέρον και συνέπειε για τα ζώα. Δεύτερον, μιλούν για την ασφάλεια των ανθρώπων όταν υπάρχουν εναλλακτικέ λύσει, γιατί θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή στι κάνε ε, των όπλων και για άλλα τεχνικά ζητήματα, τα οποία εγώ δεν τα γνωρίζω τόσο κολλά, όμω υπάρχει μεγάλο προβληματισμό ω προ αυτό. Και μετά υπάρχει και μια σκέψη ότι δεν είναι αναλογική η πρόταση ότι δεν ανταποκρίνεται στους κινδύνου που συνδέονται με το μόλιβδο και πάλι δεν είμαι ειδική, θα ήθελα να μου πείτε περισσότερα επί του θέματος για να δούμε αν ισχύει κάτι τέτοιο. Μου φαίνεται ότι δεν ε, χαίρει ε, πλήρους στήριξης αυτή η πρόταση. Κάποια από τα στοιχεία που θίγει ο Σύλλογος Κυνηγών ευσταθούν και θα ήθελα κάποιες ε, παρατηρήσεις να μου πείτε για τα όσα έθιξα. Μετά υπάρχει ένα προβληματισμό κατά πόσο υπάρχει τόσο μεγάλη συνέπεια για το περιβάλλον και για την υγεία. Θα ήθελα να μου δώσετε περισσότερα στοιχεία ω προ αυτό. Μπορώ να σα πω όμω, συνάδελφοι, ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει γύρει μεγάλες ανησυχίες ε, στους κυνηγούς που δεν συνηθίζουν να έρχονται σε επαφή ε, με το γραφείο μου. Ασχολούνται με τα δικά του οι άνθρωποι, αλλά εδώ θεωρούν ότι πρόκειται για κάτι υπερβολικό και ανάρμοστο. Και θέλω εγώ να βρω τη σωστή ισορροπία ανάμεσα ε, στα συμφέροντά τους ε, και στις επιπτώσεις για την υγεία και το περιβάλλον που αναφέρθηκαν. Διαρωτώ με κατά πόσο είναι αναλογική λοιπόν αυτή η πρόταση. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Τροπή να απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα, καθώς και στο ότι θεωρούσε ότι θα είχε περάσει από την Επιτροπή μέχρι τώρα, αλλά είναι σαφές ότι κάπου παρεμποδίζεται. Δεν είναι δηλαδή μόνο η κυνηγοί στη χώρα μου, αλλά και σε άλλες χώρες που διαμαρτύρονται. Ο κύριος Σαχίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για μα, καθώς ο ΠΟΗ αναφέρει ότι δεν υπάρχουν ασφαλή επίπεδα μολύβδου, είναι επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, για τα ζώα και για το περιβάλλον. Ελπίζω λοιπόν να μην αποδυναμωθεί αυτή η πρόταση επιτροπή από τα λόμπι των κυνηγών. Οι υγροβιότοποι είναι πολύ σημαντικοί για εκατοντάδη είδη πτηνών και άλλων ε, ε, ζώων Και υπάρχει σοβαρή μόλυνση από τον μόλυβδο που διαχέεται στο περιβάλλον ε, μέσω του κυνηγιού. Η ε, κατανάλωση τέτοιου μολύβδου από τα ε, πτηνά οδηγεί με τη σειρά τους σε άλλες δευτερογενείς πηγές ρήπανσης, δηλητηρίασης και ούτω καθεξής. Και αυτό επηρεάζει και το πόσιμο νερό πολλές φορές. και υπάρχουν τέτοιες ε, καταγγελίες ε, για ύπαρξη και ρήπανση μολύβδου ε, σε υγροβιότοπους. Βλέπουμε ότι έχουμε 1.400 έως 1.800 τόνους μολύβδου κάθε χρόνο και έχουμε ακόμα περισσότερους τόνους μολύβδου που έχει να κάνει με την αθλητική σκοποβολή κάθε χρόνο. Πρέπει λοιπόν να απαγορευτούν και στους υγροβιοτόπους αλλά και ε, σε, στις ε, χερσαίες περιοχές. Διερωτώ με ποιος παρεμποδίζει το έργο αυτής της Επιτροπής, γιατί φαίνεται ότι δεν προχωρά το έργο της. Κυρία Ντάλη, για την ίδια πολιτική ομάδα, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δώστε μου δύο λεπτά για να σα παρουσιάσω τι δικέ μου ανησυχίε, Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση και κατανοώ ότι υπάρχουν κίνδυνοι για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που απορρέουν από τα βλήματα μολύβδου στου υγροβιοτόπους και γύρω από αυτού. Συμφωνώ λοιπόν με την επιχειρηματολογία της Κομισιόν, όμως θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τα ίδια σας τα λόγια στην παράγραφο 29, όπου λέτε ότι υπάρχει ανάγκη ε, το μέτρο να είναι και αποτελεσματικό, αλλά και απλό και δίκαιο. Και εξηγούμε. Προέρχομαι από τη Μάλτα, μια πολύ μικρή χώρα, ένα μικρό νησί στη Μεσόγειο, περικλείεται από νερό προφανώς. Και εκεί υπάρχουμε και κυνηγού, έχουμε και κυνηγού, ε, ε, σκοπευτές που ασχολούνται με σκοποβολή για λόγους ψυχολογίας και τα καθεξής. Για μένα λοιπόν οι υγροβιότοποι Φυσικά και θα πρέπει να συνεχίσουμε να προστατεύονται, δεν υπάρχει ζήτημα. Αυτό έλεγα στην αρχή. Αλλά το βασικό ζήτημα εδώ είναι ο ορισμό του υγροβιότυπου που ε, χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί στο σχέδιο κανονισμού αναφέρεται σαφώ ότι βασίζεστε στον ορισμό του υγροβιοτόπου που χρησιμοποιείται στη Σύμβαση 1971. Και εκεί περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων περιοχές νερού, είτε πρόκειται για θαλασσινό νερό, ε, γλυκό νερό, αρκεί να μην ε, ε, υπερβαίνει τα έξι μέτρα η παλήρια και άμποτη. Ο ορισμός αυτός λοιπόν θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο στα μικρά νησιά και στη Μάλτα. Δυστυχώς, ο κανονισμός δεν λαμβάνει υπόψη ε, τις ιδιαιτερότητες επιμέρους κρατών μελών. Ε, δεν επιτρέπεται το κυνήγι στους οικογραφιότοπους ούτε στα θαλάσσια, νερά, στα θαλάσσια ύδατα ε, κάτω των 6 μέτρων. Όμως, η πρόταση της Επιτροπής σημαίνει ότι η ζώνη ανάσχεσης θα αφορά τελικά το μεγαλύτερο κομμάτι των ακτών των νησιών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος των νησιών ή το οικοδομημένο περιβάλλον δεν ξέρω πώς προτίθεται να λύσει αυτό το ζήτημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί σίγουρα δεν πρόκειται να καλύπτει όλα τα κρατημέλη με τον ίδιο τρόπο αυτή η πρόταση. Και αυτό με φέρνει σε άλλα ζητήματα. Στο προσχέδιο η Επιτροπή αναφέρει ότι υπάρχουν άλλες εναλλακτικέ λύσεις, ε, τεχνητά βιώσιμες ε, και προσιτές οικονομικά. Άλλοι μου έχουν πει ότι δίνει την εντύπωση αυτό το, αυτή η διατύπωση ότι με άλλα υφιστάμενα μέσα μπορούμε να λύσουμε αυτό το ζήτημα και μου είπαν ότι δεν ισχύει αυτό. Εσείς τι ανταπαντάτε. Άλλο ισχυρισμό, ότι υπάρχει πρόθεση εδώ να απαγορεύσουμε την, ε, την αθλητική σκοποβολή. Ε, παρότι οι περισσότερες, τα περισσότερα βλήματα μολύβδου που ε, χρησιμοποιούνται ανακτώνται και επαναχρησιμοποιούνται. Εσείς τι λέτε ως προς αυτό. Και τέλος, η οπλοκα... κάτοχοι όπλων μάλλον για εθελοντικούς λόγους λένε ότι η αλλαγή προς άλλα υλικά που δεν είναι μολύβδου ε, τελικά θα πλήξει το συνολικό τομέα και θα τον καταστήσει παροχημένο. Ποιες είναι οι δικές απαντήσεις. Κύριε Στόρμπαλς, για την ομάδα Ρενιού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια πρώτη παρατήρηση εγώ να σας πω ότι έχω ε, μία, ένα τέτοιο κυνηγητικό όπλο διαμετρήματος 12 χιλιοστών. Και όπως λέω πάντα, δεν μοιράζομαι τη γυναίκα μου, ούτε σας δίνω το σκύλο μου, αλλά μπορώ να σας δώσω την καραμπίνα μου. Τώρα, υπάρχει μια παλαιά συμφωνία σε ό,τι έχει να κάνει με τα, το κυνήγι πτηνών, με την Ευρωπαϊκό Σύλλογο Κυνηγών και τη σταδιακή κατάργηση των ε, εμβλημάτων μολύβδου στους σκορβιότοπους. Εδώ λοιπόν συμφωνούμε, δεν υπάρχει λόγος να το ε, ξανασυζητήσουμε. Όμως, Εάν ε, θέλω να κυνηγήσω φασιανούς ε, στα φιλανδικά δάση και χρησιμοποιήσω ε, κυνηγητικό όπλο με χάλιβα, παρότι θεωρώ ότι είμαι καλός στο σημάδι, βέβαια άλλοι μπορούν να διαφωνούν, κάποια βλήματα σίγουρα θα πετύχουν τα δέντρα. Αυτό σημαίνει ότι ε, θα πλήξουμε έτσι τη δεντροκομία, την ε, υλοτομία. Κανεί δεν θα αγοράσει αυτά τα δέντρα. Για πλευρά επιτροπή, λοιπόν, θα πρέπει να δούμε αν πώς επιτρέπεται ε, ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση μολύβδου όταν ο μόλυβδος δεν δημιουργεί τέτοια ζημία όσο στους υγροβιοτόπους. Αυτό θα ήταν μια καλή συμβαστική λύση όπου όλοι, την οποία όλοι οι σόφρονες θα μπορούσαν να αποδεχθούν. Ευχαριστώ κύριε Τόρμπαλ. Εκ μέρους της ID ο κύριος Χακαραένα. Kiitos puheenjohtaja. Lyijy on paras materiaali eettiseen metsästykseen ja urheiluun. Ευχαριστώ. Ο, ο μόλιβδος είναι το ένα υλικό που πείτε για ε, την σκοποβολή και το κυνήγι. Υπάρχουν άλλα υλικά που είναι πιο ε, ακριβά ή δημιουργούν άλλα προβλήματα. Η μελέτη οικονομικού αντικτύπου λαμβάνει υπόψη εδώ μόνο το κυνήγι, ενώ με την πρόταση αυτή θα επηρεαστούν και άλλες ε, μορφές σκοποβολής. Εξετάσαμε μόνο τους υγροβιοτόπους. Δεν πρέπει να εξετάζουμε αυθαίρετα τις διάφορες ε, ζώνες ανάσχεσης. Οι περιορισμοί θα πρέπει να αφορούν περισσότερο ε, τα λιμνάζοντα νερά και έτσι να είναι αναλογική η πρόταση σε σχέση με πιθανούς κινδύνους. Μια τέτοια απαγόρευση υπάρχει στα περισσότερα κράτη-μέλη. τέτοιου είδους απαγόρευση θα δυσκολέψει πάρα πολύ τις μεγάλες χώρες να ε, ελέγξουν ε, αυτές τις ε, ζώνες απαγόρευσης. Τα παιδεία σκοποβολής θα πρέπει να μείνουν εκτός αυτών των περιορισμών, γιατί η ζημιά αυτή μπορεί να καλυφθεί με άλλους τρόπους μπορεί να αλλάξει ο προσδιορισμός των ζωνών και τα άλλα υλικά έχουν κινδύνους. Αυτό δεν το λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα βλήματα χάλιβα έχουν απαγορευθεί ε, σε πεδία σκοποβολής για περιβαλλοντικούς λόγους. Και δεν αξιολογείται ε, ο αντίκτυπος αυτών των απαγορεύσεων εδώ. Υπάρχει κι άλλη πρόταση ε, ιδεολογική ευρωπαϊκού ε, προσανατολισμού, ο τελικός στόχος είναι η πλήρης απαγόρευση ε, κατοχής όπλων από τους πολίτες. Και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουμε αυτή την ε, απαγόρευση. Ποιος θα αποζημιώσει τον κάτοχο ενό, ενός όπλου που πλέον δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει. Το κόστος της παρακολούθησης και εφαρμογής του νόπου θα είναι αστρονομικό. και η απαγόρευση κατοχής βλημάτων μολύβδου θα είναι πολύ δύσκολη. Δεν μπορεί να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιες απαγορεύσεις ε, στην ε, νομοθεσία των κρατών μελών, είτε θα είναι ε, μία άστοχη νομοθεσία χωρίς περιοχόμενο ή θα πρέπει τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν αυτή τη νομοθεσία, που μπορεί να είναι αντισταγματικό για την επιμέρους χώρα. Όπως και να έχει, δυσκολεύει τη ζωή των ε, κυνηγών, ακόμα και την ε, ίδια τη βιομηχανία, τους λόγους κυνηγών, ε, την οπλοβιομηχανία, τους αξιωματούχους, ακόμα και το στρατό. Δεν ξέρω, είναι αυτό αναλογικό ε, κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ευχαριστώ κύριος Φιόκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. θα πω κάτι για τους συναδέλφους δεν το γνωρίζουν. Ο Μόλιβδος χρειάζεται να έχει την ε, ε, εξουσιοδότηση του ρίτς, απαγορεύεται να χρησιμοποιείται στην αλληλεία, στο κυνήγι, κοντά στους ε, υδροβιοτόπους. Όσον αφορά την εξουσιοδότηση από το ρίτς, Ξέρουμε ότι είναι στον κατάλογο των ε, ουσιών εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων που βρίσκεται στην Ευρώπη ε, σε πολλά προϊόντα. Προσπαθήσαμε να τον βγάλουμε από τις μπαταρίες πρώτα απ' όλα. Επίσης, ξέρουμε ότι 80% του μολύβδου χρησιμοποιούνταν παλιά στις μπαταρίες και προσπαθήσαμε αυτό να το διορθώσουμε. Δεύτερον, θα ήθελα να επισημάνω ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορες κοινωνικονομικές μελέτες όσον αφορά το μόλυβδο, η απαγόρευση χρήσης του ως ουσία θα δημιουργήσει σε πρόβλημα κάποιες οικονομίες στην Ευρώπη. Γι' αυτό ξέρουμε ότι κάποιες ε, παραγωγή προϊόντων με μόλιβδο θα μεταφερθούν στις Τουρκία στην Κίνα. Όταν εξετάζουμε αυτές τις διαδικασίες περιορισμού χρησιμοποίησης, με μέρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρησιμοποίηση ε, ε, του μολύβδου κοντά στους υγροβιοτόπους ήμουν μέλο όλη αυτή τη διαδικασία στην ΕΠΑ. Πρέπει να πω ότι είναι, η παρά το γεγονό ότι τους προσάπτουμε πολλά, πολύ μπροστά. Λέγεται ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το κυνήγι της πάπιας ή της χίνας. Κατά διάρκεια τη κυνηγετική περίοδου για αυτά τα, για τεινά. Τέλος. Τώρα, για να προστατευτεί το, ε, η εδώ και 40 χρόνια προσπαθούν να κάνουν κάτι για να περιορίσουν τη χρήση τους τους υγροβιότοποι. Το πρόβλημα δεν είναι ο περιορισμός τους, διότι συμφωνούν οι περισσότεροι κυνηγοί αλλά διότι υπάρχει μια σευρύτατος ορισμός όσον αφορά τους ε, υγροβιότοπους και θα πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει GPS για να δει αν είναι εντός του χώρου του υγροβιότοπου ή εκτός. Τώρα, όσον αφορά τα κυνηγητικά όπλα, αν έχει κανείς τέτοιου είδους φυσίγγια στην Ιταλία, διαπράττει ποινικό δίκημα. Βλέπετε λοιπόν πόσο άδικο είναι αυτό για πολλούς πολίτες. Τελικά, όταν μιλούμε για την απαγόρευση του μολύβδου, θα πρέπει κανείς να το απαγορεύσει και από την σκοποβολή. Τι θα κάνουμε. Και από τις ε, θα το απαγορεύσουμε και από την ε, σκοποβολή ως ε, άθλημα. Θα πάμε στους Ολυμπιακούς. Ε, πώς. Αυτή τη χρήση την έχουμε σκεφτεί. Επίσης, υπάρχει και θέμα ανακύκλωσης, όπως των στόχων του μολύβδου, των πλαστικού. Όλα αυτά είναι πολύ καλά για το περιβάλλον. Και τώρα μας λένε ότι δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. για την ε, ανακύκλωση και για τη χρησιμοποίηση των κυκλωμένου ε, μολύβδου παίρνει κανείς για το 900 ευρώ. Αυτή την δραστηριότητα την απαγορεύσουμε. Πιστεύω ότι χρήσιμο χρήση του είναι πολύ κακή, το λένε όλες οι επιστημονικές μελέτες, κυρίως για τα παιδιά, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ελέγξουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δεδομένα εδώ και 40 χρόνια επιστημονικά που μας λένε πώς μπορούμε να ελέγξουμε το προϊόν αυτό. Θα ήθελα λοιπόν η Επιτροπή στην προσέγγιση της να είναι ε, ε, να, μελετήσει όλα αυτά τα στοιχεία για να μπορέσει να κάνει μια περιστατωμένη μελέτη. Διαφορετικά όλα αυτά τα θετικά στοιχεία τα βάζουμε στο περιθώριο. Επίσης, ξέρουμε ότι η απαγόρευση ε, χρήσης μολύβδου είναι κάτι το οποίο στις μεσογειακές περιοχές θα βλάψει τους κυνηγού. που είναι φτωχοί. Όλα αυτά επιβάλλονται από τις Βρυξέλλες. Αυτή είναι η υποψή τους και αυτό δεν θέλουμε να το κάνουμε εμείς. Πιστεύω ότι έχουμε το ειδικό καθήκον να δείξουμε σε όλους ότι η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί για τους πολίτες της και όχι το αντίθετο. Σας ευχαριστούμε κύριε Γιώτη. Η κυρία Νόβακ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, το να μπορέσουμε να ελέγξουμε τον ε, περιεκτικότητα σε μόλιβδο των πολεμοφοδίων Καλό είναι, αλλά δεν νομίζω ότι η προσέγγιση τη Επιτροπής λύνει πλήρως το πρόβλημα, τουλάχιστον όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για ποιο λόγο, διότι οι προτάσει που κάνει δεν ελέγχει και δεν περιορίζει ε, την ε, περιεκτικότητα μολύβδου στα φυσίγγια και στα σφαιρίδια. Ο κατασκευαστής είναι αυτός ο οποίος ξέρει τις λεπτομέρειες και μπορεί να ε, αντικαταστήσει στα πλαίσια των δυνατοτήτων μόλιβδο με κάποιο άλλο εκρηκτικό υλικό. Ο τελικός χρήστης δεν έχει αυτές τις τελικές γνώσεις. Θα πρέπει λοιπόν μόνο όσος, μόνο όποιος γνωρίζει την τεχνική πλευρά του όλου να ασχοληθεί κατά πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, δεν αναφέρεται πότε τεχνικά μέτρα που προβλέπονται θα τεθούν σε εφαρμογή. Η ερώτησή μου είναι, οι κατασκευαστές ε, έχουν αναλάβει δεσμεύσεις να αντικαταστήσουν τον μόλιβδο ή όλα πέφτουν στο νόμο των τελικών χρηστών. Ευχαριστώ. Ε, dziękuję panie przewodniczący. Ε, ołów jest wyjątkowo toksycznym metalem ciężkim. W naturze nie ulega rozkładowi, odkłada się i kumuluje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 Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώ πρέπει να διαπιστώσω ότι η παρουσίαση που έκανε η Κομισιόν για την πρόταση αυτή φαίνεται επιπόλαια. Δείχνει ε, μια ε, πρόδειλη αποστροφή προς το κυνήγι. Βασίζει την πρότασή της σε υποτιθέμενα στοιχεία όπως είναι ο θάνατος πάνω από ένα εκατομμύριο ε, πουλιών και ακούσαμε ότι η ποσότητα του μολύβδου που διαχέεται είναι 18-20 τόνοι ο συνάδελφος προηγουμένως είπε 500 τόνοι. Ο καθένας δίνει ό,τι νούμερο του έρχεται στο κεφάλι, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Αν αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό ξεκινώντας από μια ιδεολογική αποστροφή προς το κυνήγι, δεν πάμε πουθενά. Ε, πρόκειται για μια ιδεολογική αποστροφή απέναντι σε μια νόμιμη δραστηριότητα που ρυθμίζεται και καλύπτεται από την νομοθεσία. Αντίθετα, αν προχωρήσουμε σε μια αξιολόγηση της κατάστασης αυτής, ε, ο αριθμός των πουλιών που χάνονται δεν σχετίζεται με την κοινωνική δραστηριότητα, αλλά με την καταστροφή των υγροβιότοπων. Στην Ευρώπη υπάρχουν ακόμα τέτοιοι βιότοποι που τα ε, υδρόβια πουλιά ε, μπορούν να ζήσουν και να πολλαπλασιαστούν, και αυτό δεν, γίνεται, δεν, δεν, ε, κινδυνεύει από τη δραστηριότητα των κυνηγών. Ε, αντίθετα, οι υγροβιότοποι υπάρχουν χάρη στους κυνηγούς. Έχουμε ε, μπορέσει να διαπιστώσουμε με αντικειμενικές αποδείξεις ότι οι η ε, υδρόβια ε, χλωρίδα και πανίδα βρίσκεται σε συνεχή αύξηση ακριβώς χάρη στην ε, προσπάθεια διατήρησης των φυσικών υγροβιότοπων. Τώρα, αν θέλουμε να αφήσουμε κατά μέρος τις ιδεολογίες σχετικά με ε, το κυνήγι. Γιατί χρησιμοποιούνται αυτά τα πυρομαχικά που περιέχουν μόλιβδο. Γιατί ο μόλιβδος είναι ένα μαλακό και βαρύ μεταλλό που ε, παραμορφώνεται κατά την είσοδό του στο ζώο και το σκοτώνει χωρίς να προκαλεί ε, ε πόνο δεν υποφέρει το ζώο. Είναι η βαλιστική του συμπεριφορά σαφώς καλύτερη από ότι οποιοδήποτε, οποιοδήποτε άλλου μετάλλου. Και εξάλλου ε, ε, έχουν γίνει πειράματα με χρήση άλλων ε, μετάλλων όπως είναι το ε, ατσάλι παραδείγματος, ο χάλιβας που δεν παραμορφώνονται γιατί είναι πιο σκληρά και ε, τι γίνεται, ε, δέχεται αυτό το χτύπημα ε, το ζώο χωρίς να σκοτώνεται επί τόπου. Ε, το αποτέλεσμα λείπει και πάει κάπου αλλού και πεθαίνει. είναι η κατάσταση δηλαδή πολύ χειρότερη από αυτή που προκύπτει από το βλήμα μολύβδου. Τώρα, για την υγεία του ανθρώπου το πόσιμο νερό, οι σωλήνες μέσω των οποίων περνάει το πόσιμο νερό, ε, είναι από μόλιβδο, αλλά ίσως δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ε, τώρα, για, το, για την άγρια ε, πανίδα, υπάρχει ένα παθολογικό πρόβλημα που δημιουργείται από την ε, κατάποση μολύβδου από ε, τα υδρόβια πτηνά, πρέπει να σας βεβαιώσω ότι τα πουλιά αυτά τρώνε διάφορα πράγματα, αλλά δεν τρώνε μόλιβδο. Για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα που λέγεται σατουρνισμό, θα έπρεπε να ε, καταπιούν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες μόλιβδου. Είναι αδιανόητο να σκεφτεί κανείς ότι θα καταπιούν τέτοιες τεράστιες ποσότητες μολύβδου τα άγρια πτηνά. Τώρα, όσον αφορά τα αποτελέσματα που θα προκληθούν, Ήδη υπάρχουν ε, και έχουν αναφερθεί κάποιες ε, διεθνείς συμβάσεις, ε, τις οποίες έχουν υπογράψει και η Ιταλία και 20 άλλες χώρες, με σκοπό την απαγόρευση των βλημάτων μολύβδου σε ε, τέτοιους υγρότοπους που ορίζονται στα πλαίσια του δικτύου Natura 2000. Στην Ιταλία σε όλα τα μέρη που καλύπτονται από το Natura 2000 απαγορεύεται η χρήση των ε, ε, βλημάτων αυτών ακριβώς για να ελεγχθεί αν η χρήση ε, βλημάτων με άλλα μέταλλα ε, έχει πιο θετικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, σε άλλες χώρες είδαμε ότι επανήλθαν στη χρήση των βλημάτων μολύβδου ακριβώς γιατί έχουν, ε, καλύτερε, έχει καλύτερες βαλιστικές ιδιότητες από τη χρήση άλλων μετάλλων που είναι πιο ελαφρά και για να έχουν ε, την ε, ε, βαλιστική συμπεριφορά που είναι επιθυμητή, πρέπει να αυξηθεί η όθηση που δίνεται στο βλήμα. Όταν χρησιμοποιούνται λοιπόν πυρομαχικά διαφορετικά από ό,τι του, του μολύβδου, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουν όλες οι κάνες των κυνηγητικών όπλων, διότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με φορτίο ε, πυρομαχικού, ε, που είναι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται από τη χρήση του μολύβδου. Όλα αυτά θα πρέπει να ταξιολογήσει η Κομισιόν, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε λόγω ε, ιδεολογικών θεωρήσεων να ε, προχωρήσουμε σε μέτρα που να μην βασίζονται σε αντικειμενικούς λόγους, αλλά ε, διότι βασίζονται σε ένα ιδεολογικό κυνήγι, αν μπορώ να το πω έτσι, τις δραστηριότητες του κυνηγιού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ, δεν ξέρω, βλέπω τον κύριο Μπόντρα, άρα δίδω το λόγο στην κυρία Πάουλου, εκ μέρους των Πρασίνων. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ομολογώ ότι με εκπλήσουν οι συζητήσεις ε, και τα όσα ακούγονται σήμερα εδώ. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη Μάρκο Βάλστρουμ. Ήταν επίτροπος περιβάλλοντος σε μια εποχή όπου υπεγράφει αυτό το, εδώ το έγγραφο. Πρόκειται για τη συμφωνία μεταξύ της FACE και της Good Life. Μια συμφωνία δηλαδή μεταξύ του Συλλόγου Κυνηγών και του ε, Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος. Ε, είχε υπογράψει ο Ζουρμπεντ Γκρουκχάιμ από την FCE και ο Μίχαλ Ράντς. Το 2004 όλα αυτά. Σε αυτό το έγγραφο αναφέρει μια παράγραφο και τις δύο οργανώσεις, όχι μόνο την Good Life, που ζητούν και οι δύο λοιπόν τη σταδιακή κατάργηση των ευλημάτων μολύβδου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το μέτρο δυνατών όπω και να έχει πριν από το 2009. Εάν δεν κάνω λάθο, έχουμε 2020 πια. Έχουμε μια συμφωνία που συνυπέγραψε και η οργάνωση ε, κυνηγών. Και τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί ασκούν πιέσει για μια νευροτοξική ουσία που θα έπρεπε να έχει καταργηθεί εδώ και πολύ καιρό, αν με ρωτάτε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναλαμβάνει δράση για το μόλεδο αυτή τη φορά. Ε, έχει έρθει επιτέλου η ώρα να αφήσουμε αυτή την ουσία εκτός των πλέον ευάλωτων γεών που έχουμε. Αν ακούσετε τους επιστήμονες, το θέμα δεν είναι αν έχουμε 4.000 ή 5.000 τόνους μολύβδου. Δεν υπάρχουν ασφαλή επίπεδα μολύβδου. Τέλος. Δεν ξέρω πώς ελέγχουμε τον μόλυβδο που ε, διαχέεται στο περιβάλλον, στον αγροβιότοπο. Θα πάτε εσείς να το μαζέψετε με το χέρι. Τι εννοείται με τον έλεγχο ακριβώς. και πρέπει να προστατεύσουμε και τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ε, ασχολούνται με αυτό το ζήτημα. Αλλά δεν μιλούμε για μία... για έναν, ε, τον έλεγχο και τον περιορισμό ενός πληθυσμού, ενός ε, είδου. είδους. Παρακαλώ λοιπόν την Επιτροπή να απευθυνθεί στο Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εμπλακούν. Πολλά κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη απαγορεύουν την χρήση πυρομαχικών μολύβδους στους χροβιοτόπους. Πρέπει να λάβουμε δράση λοιπόν τώρα. Ευχαριστώ. κύριος ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω το εξής και εδώ δεν υπάρχει θέμα ε, διαφορετικών συγγενών. Πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι ε, κυνηγό, όχι επαγγελματία. Ξέρουμε ότι από αυτού του θέματος απέριψε μία σχετική πρόταση από μία πάρα πολύ ε, ολιγομελή ε, πολιτικό κόμμα, ολιγομελές πολιτικό κόμμα. Όλοι, όλοι, οι μεγάλοι το απέρριψαν. Και πολύ καλά. Θα ήθελα να μου πείτε πιο ένα άτομο το οποίο έχει μολυνθεί από τη, μεταξύ των κυνηγών από μόλυβδο. Έναν. Σύμφωνα με μια έκθεση της ΦΕΙΣ αναφέρεται κάτι τέτοιο. Ποιος εκπροσωπεί, εμένα δεν με εκπροσωπεί. Τώρα, ο μόλυβδος δεν χρησιμοποιείται μόνο για το κυνήγι χρησιμοποιείται για τη σκοποβολή, στα αθλήματα. Και πρέπει να σας πω, οι περισσότεροι ε, αθλητικοί όμιλοι και ομάδες σήμερα έχουν συστήματα περί συλλογής του μολύβδου. Υπάρχουν τέτοια συστήματα τα οποία επιτρέπουν τη συλλογή του μολύβδου και την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Επίσης, πρόκειται για ένα επιδεολογικό θέμα. Και εδώ δεν δίδεται ένα αμφιβόλο ο μόλυβδος ο οποίος είναι παρόν παντού, στα σπίτια μας, στα δημόσια κτίρια. Είναι λοιπόν το θέμα ιδεολογικό. Στην ε, προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου ασχοληθήκαμε με τα όπλα. Τώρα ασχολούμαστε με το μόλιβδο. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά. Ξέρετε πόσες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη ζουν από την ε, χρησιμοποίηση τέτοιων στην Πορτογαλία, στην ε, ε, Γερμανία, σε άλλες χώρες. Ξέρετε πόσες θέσεις εργασίας ενέχονται εδώ. Ποιος συμμετείχε σε αυτή τη μελέτη που έχουμε εδώ πέρα μπροστά μας πόσα άτομα που έχουν σχέση με την ε, βιομηχανία, με το κυνήγι, που έχουν σχέση με τις κυβερνήσεις μέσω των ε, θεσμικών οργάνων που είναι υπεύθυνα για τη ρύθμιση του κυνήγιου έχουν συμμετάσχει. Επίσης, πώς συμπεριφέρεται ο μόλιβδος που είναι μέσα στα φυσίγγια που χρησιμοποιούνται, τι μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς. Γιατί Ξέρουμε πώς ε, συμπεριφέρεται το φυσίγγι, το σφαιρίδιο στο κυνηγητικό όπλο. Υπάρχει κάποιο άλλο μέταλλο, κάποια άλλη εκρηκτική ουσία που μπορεί να κάνει ό,τι κάνει ο μόλυβδος. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να ανοίξουν τα μάτια τους στα, στην, πραγματική, στην πραγματικότητα, στη λογική σήμερα. Τα περισσότερα άτομα που ζουν σε αστικές περιοχές πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλλουν το δικό τους το πρότυπο στον υπόλοιπο κόσμο. Στις περισσότερες χώρες μας τα περισσότερα άτομα ζουν στην ύπεθρο και τα άτομα που ζουν στις περιοχές έχουν τη δική τους πραγματικότητα. Τα άτομα λοιπόν τα οποία θα αποδεχθούν αυτού του είδους τα μέτρα δεν πρέπει να τα καταλάβουν πριν να τα αποδεχθούν. Όταν λοιπόν μιλούμε για μόλιβδο, θα ήθελα να μου δώσετε επιστημονικές εξηγήσεις και ευρήματα και όχι να βασίζετε σε ιδεολογικά θέματα. Και θα τελειώσω όπως άρχισε. Θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να βρει ποιοι συμμετείχαν στη σύνταξη αυτή της μελέτης. Υπάρχουν επιστήμονες ειδικοί που έχουν συμμετάσχει. Θέλω να μου απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μέλο. Ήρθε και ο κύριος Μπόντα από την ΙΣΙΑΡ, του δίνουμε αμέσως το λόγο. You know, usually, as you know, I Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, ε, είμαι εδώ συνήθω ε, για να υπερασπίζω με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενάντια στον ριζοσπαστισμό, ριζοσπαστικότητα όλων ημών. Τώρα όμως νομίζω ότι η Κομισιόν το παράκανε. Δεν είμαι ούτε κυνηγό ούτε ψαράς. Αλλά τρώω το κυνηγί τρώω και ψάρια και γλυκού και θαλασσινού νερού και είμαι υγιής. Δεν έχω πάει στο γιατρό ούτε μια φορά στη ζωή μου. Νομίζω ότι είναι κάπως ιστερική αυτή η αντίδραση, η δαιμονοποίηση του μόλιβδου, η δαιμονοποίηση των ε, κυνηγών και δεν καταλαβαίνω. Είμαι και ο, ε, ερασιτέχνης ορνηθολόγος εγώ είμαι υπέρ της απαγόρευσης και είμαι ε, και έχουμε στη χώρα μου απαγόρευση στους υγρότοπους. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί η Κομισιόν το πάει τόσο μακριά. Μετά από αυτή τη συμβαστική λύση, ε, σύμφωνα με την οποία όλοι στις χώρες μας και οι κυνηγοί και οι λάτρεις των πουλιών μπορούν να συνεπάρξουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Κομισιόν αποφάσισε να προχωρήσει τόσο πολύ με αυτές τις συστάσεις, μειώνοντας την μεταβατική περίοδο και αποφασίζοντας για νέες ε, προστατευόμενες ε, ζώνες και αυτόματα έτσι ε, ποινικοποιώντα το κυνήγι με τη χρήση αυτού του τόσο διευρυμένου ορισμού των υγρότοπων. Τα μέτρα αυτά που προτείνονται δεν ε, αναφέρουν ε, κατά πόσον ε, η απαγόρευση αυτή αφορά την χρήση αυτών των πυρομαχικών από το στρατό ή την αστυνομία. Αν ένας αστυνομικός κυνηγάει ένα κακοποιό και υπάρχει μια λίμνη εκεί γύρω, δεν μπορεί να ενεργήσει κατά την άποψη της Κομισιόν. Όσον αφορά την πλήρη απαγόρευση του μολύβδου, γιατί η την αστυνομια αν ειναι αστυνομικος κυνηγαει ενα κακοποιο και υπαρχει μια λιμνη εκει γυρω δεν θεωρεί ε, δεν λαμβάνει υπόψη ένα περιορισμό που να πηγαίνει παραπέρα. Γιατί μάλλον προτείνει ένα περιορισμό που ξεπερνάει τη συμβαστική λύση που είχε βρεθεί. Και κάτι άλλο. Στη χώρα μου έχουμε 400.000 κυνηγούς και περίπου άλλους τόσους ψαράδες. Και δεν είναι όπως ε, στην Ολλανδία που έχετε αυτούς τους εκατομμυριούχους που κυνηγάνε επάπιες. Στη χώρα μου οι κυνηγοί είναι οι, οι απλοί φτωχοί άνθρωποι που ζουν στην Ήπεθρο. Αν τους αφαιρέσετε αυτό το χόμπι δεν είναι ε, σε θέση να βρούνε άλλον εξοπλισμό. Ούτε οι κυνηγοί, ούτε οι ψαράδες, αν προχωρήσετε σε πλήρη απαγόρευση. Πρόκειται για μια συνταγή για το πώς ένα εκατομμύριο περίπου πολίτες στη χώρα μου θα στραφούν ενάντια στην Κομισιόν, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν πρόκειται να καταλάβουν γιατί το κάνετε αυτό και εγώ σαν ορνηθολόγος μπορώ να σας πω ότι δεν θα προστατεύσετε κανένα πτηνό με τον τρόπο αυτό. Τα πτηνά αναπτύσσονται μια χαρά στους υγρότοπους μας και μπορώ να σας πω ότι δεν χρειάζονται τέτοιες δραματικές κινήσεις. Τελείωσε ο γύρο των ομιλητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριο Πετινέλη, εκ μέρου Κομισιόν, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για μια ιδιαίτερα πλούσια ανταλλαγή απόψεων. Θα ξεκινήσω με το ερώτημα του κυρίου Λίζε, που ζήτησε να την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει μια ισορροπημένη λύση, να μην υπερβάλλει και συμφωνούμε απολύτως. Αυτό που παρουσιάσαμε σήμερα και μπορώ να σας πω και τώρα είναι η πρόταση για την απαγόρευση βλημάτων μολύβδου στους υγροτόπους. Για τις άλλες πιθανούς περιορισμούς βρισκόμαστε σε πολύ αρχικά στάδια της διαδικασίας. Δεν υπάρχει πρόταση της Επιτροπής, ούτε μελέτη της ΕΚΑ. Απλώς ζητήσαμε από την ΕΚΑ να προετοιμάσει το φάκελο, όπως λέμε. Δεν ξέρουμε λοιπόν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Όλες μου οι απαντήσεις λοιπόν θα περιοριστούν στο πρώτο τμήμα στην πρόταση για την ε, απαγόρευση βλημάτων μολύβδου στους υγροτόπους, το οποίο αυτή τη στιγμή συζητάται με τα κρατη Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν πρόκειται για μία υπερβολική πρόταση, είναι ισορροπημένη. Και αυτό γιατί έχει υπάρξει ε, ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη και εκτεταμένη συζήτηση που τώρα γίνεται με εκπροσώπους των κρατών μελών. Αλλά προηγουμένως υπήρχε μια ευρεία δημόσια διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν και σύλλογοι κυνηγών και πολλοί ευρωβουλευτές... Ε, γνωρίζουν ότι μεταξύ της ε, Build Life και του κυνηγετικού συλλόγου, του Ευρωπαϊκού Συλλόγου, υπήρχε συμφωνία πριν αρκετά χρόνια για την ε, απαγόρευση της χρήσης μολύβδου στους υγροτόπους. Απλώς λοιπόν εμείς εφαρμόζουμε αυτό που είχαν αποφασίσει να κάνουν και οι κυνηγοί πριν από αρκετά χρόνια. Για τα ζητήματα της κυρίας Μαγκίνε. ευχαριστώ αρχικά πολύ για την επικοδοματική ανταλλαγή απόψεων που έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Για τον ορισμό των υγροτόπων, δεν ε, θέλουμε εδώ να επινοήσουμε από την αρχή τον ε, τροχό. Υπάρχει σύμβαση που έχει υπογραφεί από όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχει η Ράμσακ, Ραμσάρ με τον ορισμό των υγροτόπων που έχει υπογραφεί από όλα τα κρατημέλη και μια άλλη σύμβαση για την καλύτερη ζωή, Better Life, που έχουν υπογράψει μόνο 23 από τους 27. Ήδη υπάρχει λοιπόν ένας διεθνώς αναγνωρισμένος ε, ορισμός, τον οποίο έχουν υπογράψει τα κρατημέλη και εμείς αυτόν θέλουμε να αξιοποιήσουμε. γιατί τη ζώνη ανάσχεση τώρα, Ζώνε ανάσχεση. Πρέπει να βρούμε μία λύση, ακόμα εκρεμεί αυτό το ζήτημα. Η τρέχουσα πρόταση είναι... Ε, να καταλήξουμε σε έναν αριθμό μέτρων, για παράδειγμα 200 μέτρα, κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι τόσο σαφείς γιατί κάποιες φορές λέμε, έχουμε διατυπώσεις όπως ε, περιοχές κοντά, ας πούμε. Και αυτό είναι δύσκολο να το προσδιορίσουμε. Προτείνουμε εμείς λοιπόν να δώσουμε έναν σαφή και πολύ ρητό αριθμό. Ε, βεβαίως αν υπάρχει διαφορετική πλειοψηφία θα προσαρμόσουμε την πρόταση. Και για το επαρκές χρονικό διάστημα ακόμα συζητείται αυτό. Ε, δεν έχει υπάρξει συμφωνία. Ξέρουμε ότι οι Ιρλανδοί κυνηγοί έχουν διαφορετική θέση από τους συλλόγους κυνηγών των ε, χωρών ε, τους. Δεν ξέρουμε γιατί, αλλά διευκρινίζουμε ότι σήμερα δεν μιλούμε για τις σφαίρες, μόνο για τα βλήματα. Κάτι τελείως διαφορετικό. Κάποιος από τους σοσιαλιστές έθεσε ένα ερώτημα, δεν κατανόησα το όνομα. Εάν υπάρχει κάποιος που παρεμποδίζει τη διαδικασία στην Επιτροπή. Όχι, δεν υπάρχει. Κάθε φορά που τίθεται το ζήτημα στην Επιτροπή γίνεται μία σε βάθος ε, και πολύ ζωντανή συζήτηση, όπως έγινε και σήμερα εδώ στο Κοινοβούλιο. Κανείς λοιπόν δεν εμποδίζει ε, τη διαδικασία, συνεχίζονται οι συζητήσεις. Η κυρία Ντάλη τώρα. Είπατε ότι πρέπει να έχουμε έναν απλό και δίκαιο κανονισμό. Ναι, για να γίνει απλός, προτείνουμε και εμείς να έχουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό μέτρων για τη ζώνη ανάσχεσης. Τώρα, για το πόσο είναι δίκαιη η πρόταση. Θεωρούμε ότι είναι η πρότασή μας κατανοούμε ότι σε μία συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή της Μάλτας, μπορεί να υπάρχουν ε, ορισμένες δυσκολίες. Εάν ε, οι εκπρόσωποι της Μάλτας έχουν κάτι συγκεκριμένο να προτείνουν, φυσικά να τους ακούσουμε. Αλλά εμείς θέλουμε προτάσεις για λύση, όχι μόνο κριτική. Τώρα, εναλλακτικές λύσεις. Στη μελέτη της ΕΚΑ, που έχει αξιολογηθεί από τις δύο επιτροπές και την Επιστημονική Επιτροπή και την Επιτροπή για τις ε, οικονομικες Επιπτώσεις. Αναφέρεται ρητός λοιπόν ότι υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις, οι οποίες βεβαίω ενέχουν ένα κόστος. Υπάρχει μια εκτίμηση στη μελέτη της ΕΚΑ. Αναφέρεται ένα επιπλέον κόστος 25 ευρώ το χρόνο ανακυνηγό Και μετά υπάρχει και ένα επιπρόσθετο κόστος για τους κυνηγού αυτούς που θα πρέπει να προσαρμόσουν τα όπλα τους. Για την αθλητική σκοποβολή, ναι, εδώ υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, είναι ακόμα ανοιχτή η συζήτηση. Πρέπει να βρεθεί μια συγκεκριμένη λύση εδώ για, την, ε, για τους λόγους, ε, για τη χρήση όπλων, τέτοιων βλημάτων για αθλητικούς λόγους. Για Κανάινεν, ε, μιλήσατε και πάλι για τον ορισμό ε, των υγροτόπων. Υπάρχει, όπως είπα, ο ορισμός Ράμσαρ. Υπήρξαν και άλλες προτάσεις ε, να εξαιρεθούν, για παράδειγμα, οι τυρφώνες από τον ορισμό των υγροτόπων. Αλλά δεν υπάρχει πλειοψηφία που να στηρίζει αυτή την πρόταση. Γιατί εμείς πάντα πρέπει να πετύχουμε πλειοψηφία και στην Επιτροπή τα περισσότερα κράτη-μέλη στρέφονται προς την υιοθέτηση του ορισμού Ράμσαρ. Για το ερώτημα του κυρίου Φιόκη. Ο μόλυβδος στις μπαταρίες. Νομίζω ότι δεν ε, είναι σωστή εδώ η σύγκριση, γιατί πρόκειται για μια τελείως διαφορετική διαδικασία. Ο μόλιβδος που περιέχεται σε, στις μπαταρίες ε, αποτελεί τμήμα ενό τελείως κλειστού κυκλώματος. Δεν ε, απελευθερώνεται ε, στο περιβάλλον, εκτός και αν υπάρξει λαθασμένη και παράνομη χρήση, γιατί κάποιοι δεν σέβονται τον νόμο. Αλλά κατά τα άλλα δεν υπάρχει λόγος σύγκρισης, πρόκειται για τελείως, κάτι τελείως διαφορετικό. Απάντησα προηγουμένως για τον ορισμό των υγροτόπων, μετά για την εφαρμογή του νόμου στην Ιταλία. Φυσικά κάθε κράτος μέλος, ε, εάν υιοθετηθεί ο κανονισμός, θα πρέπει να υιοθετήσουν αναλογικά μέτρα για την εφαρμογή του νόμου. Δεν και αυτό στις Βρυξέλλες, να αποφασίσει δηλαδή πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος σε κάθε χώρα. Αυτό το αποφασίζουν τα κράτη-μέλη. Ο κύριος Φιώκη επίσης μίλησε για την αγωνιστική σκοποβολή. Ναι, κατανοούμε ότι υπάρχει ζήτημα εδώ και είμαστε ανοιχτοί για να βρεθεί λύση. Τώρα, για τα γραφειοκρατικά μέτρα που παίρνουν οι Βρυξέλλες. Τώρα εδώ δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τέτοια μέτρα. Γιατί Πρώτα απ' όλα πρέπει να ψηφιστούν τα μέτρα από την Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν τα κράτη-μέλη, και μετά μπορεί να υιοθετηθεί μόνο εάν Κοινοβούλιο και Συμβούλιο δεν φέρουν αντίρρηση. Σε περίπτωση που είτε το Συμβούλιο είτε το Κοινοβούλιο ε, φέρουν αντίρρηση, δεν υιοθετούνται τα μέτρα. Επομένω, όλη αυτή η δικασία βρίσκεται στα χέρια των δημοκρατικών θεσμικών οργάνων, όχι των γραφειοκρατών. Οι γραφειοκράτες κάνουν την προπαρασκευαστική εργασία και μετά τα δημοκρατικά θεσμικά όργανα αποφασίζουν. Για τους κατασκευαστές και αν συμμετέχουν. Ε, βεβαίως, είχαμε δύο διαδικασίες ευρείας δημόσιας διαβούλευσης και υπήρξε και σεμινάριο εδώ στις Βρυξέλλες το Φεβρουάριο 2019 όπου όλα τα κράτη-μέλη είχαν προσβληθεί και είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις απόψεις τους. Συμμετείχαν και οι εκπρόσωποι των κυνηγών, των ε, φιλοπεριβαλλοντικών ΜΚΟ κλπ. Κυρία Σπούρεκ, υπάρχει κίνδυνος ο κανονισμός να αποδυναμωθεί από τα κράτη-μέλη. Στο ευρωπαϊκό σύστημα το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υιοθετούν τους κανονισμούς και μετά τα κράτη-μέλη οφείλουν να, τις, ε, να εφαρμόσουν την νομοθεσία. Ιδάλλως ξεκινά μια διαδικασία επί παραβάση. Πρώτα απ' όλα όμως τα κράτη-μέλη ε, έχουν και φέρουν την ευθύνη εφαρμογή της νομοθεσίας. Και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διαδικασία επί παραβάση είναι πραγματικά λύση ε, ανάγκης, η έσχατη λύση μάλλον. Θα απαντήσω στα τελικά στον κύριο Λαντσίνη. Αξιότιμε κύριε Λαντσίνη, ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει καμία μεροληπτική προσέγγιση απέναντι στο κυνήγι. Δεν έχει καμία σχέση με το κυνήγι η το μέτρο αυτό, όπως και άλλα επόμενα μέτρα θα αφορούν άλλα είδη πυρομαχικών που δεν χρησιμοποιούνται για το κυνήγι. Μιλάμε εδώ για τη χημεία και για το μόλιβδο. Ο μόλιβδος είναι μια επικίνδυνη χημική ουσία γνωστής τοξικότητας και ένας άνθρωπος ή ένα πτηνό όταν έρχεται σε επαφή με το μόλιβο. Ε, μόλιβδο δεν έχει ε, καμία σημασία αν προέρχεται από το ο αυτός ή από από κάποια άλλη δραστηριότητα. Η βλάβη υπάρχει. Στην αρχή της παρουσίασής μου σας είπα ότι υπάρχει μεγάλη απελευθέρωση μολύβδου λόγω της χρήσης αυτών των φυσικίων και γι' αυτό η Κομισιόν προτείνει να ληφθούν αυτά τα μέτρα. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν έχουμε καμία μεροληπτική ε, στάση απέναντι στο κυνήγι όπως και απέναντι σε καμία άλλη δραστηριότητα. Όσον αφορά τώρα το θέμα της ε, βαλιστικής συμπεριφορά, η μελέτη που έκανε ο οργανισμός ΕΚΑ ε, για τα χημικά προϊόντα εξέτασε με πολλές, ε, εξέτασε λεπτομερώς το πρόβλημα αυτό. Ε, αν αντικατασταθεί ο μόλιβδος στα βλήματα αυτά, η συμπεριφορά δεν θα είναι η ίδια, αλλά σίγουρα ε, θα μπορέσουν να βρεθούν λύσεις. και πριν από πολλά χρόνια, ε, θυμάστε τι έγινε με τον αμίαντο που χρησιμοποιούταν για την μόνωση των κτηρίων. Και τελικά βρέθηκαν άλλες λύσεις, στραφήκαμε προς ε, ε, άλλα υλικά. Η αντικατάσταση αυτή προκαλεί πάντα δυσκολίες, αλλά βρίσκονται λύσεις. Θέλω λοιπόν να επαναλάβω ότι ε, η προσαρμογή Τη βαλιστική συμπεριφορά των όπλων εξετάστηκε πολύ λεπτομερώς στην Επιστημονική Επιτροπή. Επανέρχομαι στα αγγλικά τώρα. Η κυρία Πάλου μα υπενθύμισε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ συλλόγων κυνηγών και ΜΚΟ. Ισχύει, το είπα και προηγουμένω. Ε, και είναι και ένα από του λόγους που μας δυσκολεύουν κάποιε φορές να κατανοήσουμε τις διαφορετικές θέσει των κυνηγετικών συλλόγων. Γιατί έχω συναντήσει αρκετού τέτοιου συλλόγου και έχουν πολύ διαφορετικές ε, θέσει. Και είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει αυτή τη διαφορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τον κύριο Μέλλο. Ο μόλυβδος βρίσκεται παντού, είπατε. Δεν είμαι τόσο βέβαιος. Και έχουμε στοιχεία ότι ο μόλυβδος είναι επιζήμιος όπου και αν βρίσκεται. Η παρουσία του μολύβδου σε διάφορα σημεία δεν σημαίνει ότι δεν είναι επιζήμιος για την ανθρωπινή υγεία. Είναι. Γι' αυτό και ένας από τους στόχους μας είναι να περιορίσουμε το μόλυβδο όσο γίνεται περισσότερο. Όπου υπάρχει πηγή μολύβδου που απελευθερώνεται στο περιβάλλον και ε, υπάρχει έκθεση των ανθρώπων σε αυτό το ο σκοπός μας είναι να περιορίσουμε και να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Μετά, αναφέρθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπερβολική. Δεν δαιμονοποιούμε το μόλυβδο ούτε τους κυνηγού. Υπενθυμίζω, ο μόλυβδος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Αυτό είναι γεγονός, υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία. Δεν πρόκειται για καμιά δαιμονοποίηση των κυνηγών, αλλά και πάλι εγώ απαντώ με βάση την πρόταση που έχει τεθεί επιτάπητος. Βλήματα στους υγροτόπους και μόνο. Πρόκειται για κάτι αρκετά περιορισμένο και ισορροπημένο. Για τη μεταβατική περίοδο, τις ζώνες ανάσχεσης και τον ε, ορισμό των υγροτόπων, γνωρίζω ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Για αυτά τα θέματα συνεχίζονται οι συζητήσεις για να βρούμε μια καλύτερη συμβαστική λύση. Μετά για την αστυνομία. Δεν είμαι ειδικό, αλλά από ό,τι γνωρίζω δεν χρησιμοποιεί βλήματα, χρησιμοποιεί σφαίρε η αστυνομία. Οι σφαίρε δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογή αυτή τη πρόταση. Η αστυνομία όμως δεν περιέχεται στο πεδίο εφαρμογή. Αυτό μπορεί και έχουν ήδη εξαιρεθεί στο αίτημα που κάναμε προ την ΕΚΑ για άλλους πιθανούς περιορισμούς που αφορά τις σφαίρες. Γιατί η αστυνομία χρησιμοποιεί σφαίρες, πράγματι. Ελπίζω να απάντησα στα ερωτήματά σας. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συμβολή σας. Πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε κύριε Πετινέλη για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτού του θέματος. Πρέπει να σας πω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας προβλέπεται για τις 5 Μαρτίου. Λύεται η συνεδρία.